Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε, αν θέλετε. Από ό,τι έμαθα σήμερα το πρωί, τα ξεπετάξατε. Περνάμε στο σημείο 21. Καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Πιθανές λύσεις. Είναι το σχέδιο γνωμοδότης της Ιωάννα Σκριτσλεύσκα. Είναι έκθεση πρωτοβουλίας μάλιστα. Εμείς είμαστε αρμόδιοι και γνωμοδοτούν οι Επιτροπές Γυναικών Πολιτισμού και Περιφερειακών Υποθέσεων. Το λόγο έχει η συγκήτρια, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω που μου δώσετε τη δυνατότητα να παρουσιάσω σήμερα την έκθεση αυτή και όχι χθε. Σα δω συγγνώμη, αλλά χθε δεν μπορούσα να φτάσω εν γέρο στι Βρυξέλλε. Σα είχα πάντω ενημερώσει. Για άλλη μια φορά σε ευχαριστώ για τη διευθέτηση αυτήν. Προτίμασα λοιπόν την έκθεση αυτή, που όπω είπατε είναι μια έκθεση πρωτοβουλία και αναφέρεται στις δράσεις που έχουν ήδη αναλυφθεί και που έχουν ως στόχο τη βελτίωση της πολύ δύσκολης κατάστασης των νέων στην αγορά εργασίας. Προσπαθώ να δώσω κάποιες συμβουλές στα κράτη-μέλη προκειμένου να καταφέρουν να αναχαιτήσουν την αύξηση της ανεργίας, ιδίως στην ηλικιακή ομάδα των νέων. Θα ήθελα να κάνω ένα απολογισμό των όσων έχουν ήδη γίνει στα κράτη-μέλη ή να αναφερθώ επίσης και σε αυτά τα οποία πρόκειται να γίνουν πολύ σύντομα. Όσον αφορά τους νέους που δεν έχουν ακόμα ενταχθεί στην αγορά εργασίας, αλλά που πρόκειται σύντομα να ενταχθούν. Λοιπόν, από πού προκύπτει η πολύ δύσκολη αυτή η κατάσταση των νέων. Προφανώ από την οικονομική κρίση, αλλά όχι μόνο. Η κατάσταση αυτή συνδέεται με ένα πολύ κακό εθνικό σύστημα εκπαίδευση, το οποίο δεν συνάδει με τις ανάγκες αγοράς εργασία. Μέσω διαρθρωτικών λοιπόν μεταρρυθμίσεων μπορεί να θεραπευτεί η κατάσταση αυτή και όχι μόνο μέσω κατά περίπτωση μέτρων. Προτείνουμε λοιπόν εμείς να γίνουν οι απαραίτητε προσαρμογέ και να αρχίσουν να εφαρμόζονται τα κατάλληλα μέτρα. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι η βελτίωση τη απασχολησιμότητα των νέων εξαρτάται από όλη την οικονομία και από το γενικότερο οικονομικό κλίμα το οποίο μπορεί να προωθήσει την επιχειρηματικότητα. Γιατί α μην το ξεχνάμε, οι επιχειρήσει είναι αυτές οι οποίε δημιουργούν θέσεις εργασία. Ό,τι γίνεται τώρα έχει ως στόχο να βοηθήσει ε, κατά περίπτωση και κατ' με ένα κατεπήγοντα τρόπο τους νέους, προκειμένου να καταφέρουν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Οι οικονομολόγοι μας λένε όμως ότι δεν θα πρέπει με αυθαίρετο τεχνητό τρόπο να προσπαθούμε να εντάξουμε τους νέους στην αγορά εργασίας όταν δεν υπάρχουν οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας, γιατί αυτό βάλει κατά άλλων ηλικιακών ομάδων, για παράδειγμα κατά των πιο ηλικιωμένων, οι οποίοι ενδεχομένω να χάσουν τη δουλειά τους. Εγώ όταν συνομιλώ με νέους βλέπω ότι είναι πολύ δύσκολο να χρησιμοποιεί κανείς μόνο οικονομικά επιχειρήματα. Θεωρώ λοιπόν, όπως και περισσότεροι συνάδελφοι, ότι τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία έχουν δοθεί για τον στόχο της καταπολέμησης ενεργείας είναι μια ξεχωριστή γραμμή προπολογισμού από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, κονδύλι που θα πρέπει να στοχεύει προς τους νέους πτυχιούχους και στους νέους οι οποίοι βρίσκονται κάτω της ηλικίας των 30 ετών. Νομίζω ότι θα πρέπει να εγγυηθούμε επίσης την αποτελεσματικότητα των δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης και θα πρέπει να εντάξουμε επίσης και τον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή τις ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης, οι οποίες θα πρέπει να προσφέρουν μια ποιοτική, ποιοτικά προγράμματα μαθητείας και επαγγελματικής εξάσκησης, πρακτικής άσκησης μάλλον. Νομίζω επίση ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε με τα Ινστιτούτα Εκπαίδευση και με του οργανισμού υποστήριξη των νέων. Α μην ξεχνάμε επίση το ρόλο που μπορεί να δραματίσει η κοινωνία των πολιτών και οργανώσει των νέων. Όλα αυτά όμω θα πρέπει να συνδυαστούν και με μια καλύτερη υποστήριξη προ επιχειρήσει, οι οποίε επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εγγύηση για την νεολαία σε στενή συνεργασία με τι δημόσιε υπηρεσίε απασχόληση μέσω διαφόρων κινήτρων, όπως για παράδειγμα φοροαπαλλαγές, εξαίρεση από τη φορολογία και κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να προωθήσουμε περισσότερο τις επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες παρέχουν στους νέους ποιοτικά προγράμματα πρακτικής άσκησης. Για να καταπολεμήσουμε όμως την ενεργεία των νέων θα πρέπει να επικεντρωθούμε και στην επιχειρηματικότητα, στις νέες εταιρείες, στις νέες καινοτόμες εταιρείες, στις λεγόμενες start-up. Θα πρέπει να βοηθήσουμε τους νέους να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να δημιουργήσουν επιχειρήσεις, να χρησιμοποιήσουν το ταλέντο τους. Θα πρέπει να καταφέρουν οι νέοι να έχουν την απαραίτητη οικονομική υποστήριξη και θα πρέπει επίσης να έχουν τα απαραίτητα φορολογικά κίνητρα και αυτοί, ιδίω στην αρχή της επιχειρηματική τους δραστηριότητας. Οι επιχειρήσεις αυτές που δημιουργούν οι νέοι θα πρέπει να δημιουργούν και θέσεις εργασίας για άλλους νέους. Ξέρετε ότι μία περίοδος απαλλαγής από τους φόρους ήταν δύο έτη σε, στις περιόδους ευμάρειας που είχαμε στο παρελθόν. Τώρα που διανύουμε μία περίοδο οικονομικής κρίσης, νομίζω ότι θα πρέπει να επεκτείνουμε αυτή την περίοδο φοροαπαλλαγής. Να αναφερθώ επίσης στην κατάσταση στην Πολωνία όπου είχαμε πολλέ νέες πρωτοβουλίε των νέων, οι οποίοι ξεκινούσαν, στείναν τι επιχειρήσει τους, αλλά μετά από αυτή την διετή περίοδο φοροαπαλλαγή ή φορολαφρύνσεων, πολλοί νέοι αναγκάζονταν να κλείσουν την επιχείρησή τους, επειδή δεν είχαν καταφέρει να αγκιστρωθούν καλά στην αγορά. Πρέπει να σας πω επίσης ότι το ποσοστό ανεργίας είναι πάρα πολύ ψηλό ανάμεσα στους νέους. Υπάρχουν όμως και διαφορές ανάμεσα στις διάφορες περιοχές της Ευρώπης. Αλλού υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες απασχόλησης και αλλού πολύ λιγότερες. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο ένα σημαντικός παράγοντας για την καταπολέμηση ανεργίας των νέων είναι η περίφημη κινητικότητα των νέων. Υπάρχει, υπάρχουν ένα εκατομμύριο διαθέσιμες θέσεις εργασίας αυτή τη στιγμή, οι οποίες δεν καλύπτονται. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να καταφέρουμε να συντονίσουμε καλύτερα και το φαινόμενο της κινητικότητας των νέων, αλλά και τη δυνατότητα μεταφοράς των συνταξιδοτικών δικαιωμάτων. Επίσης, θα πρέπει να προωθήσουμε τις γλωσσικές δεξιότητες που συμβάλλουν στο να βρεθεί μια θέση εργασίας. Επίσης, να υποστηρίξουμε περισσότερο το δίκτυο EURES, το οποίο βοηθά τους νέους να βρουν την πρώτη τους εργασία. Ας προωθήσουμε λοιπόν περισσότερο το πρόγραμμα EURES, ας του δώσουμε μεγαλύτερη προβολή και ας καταστήσουμε την εργασία του πιο αποτελεσματική. Ξέρετε ότι πολλοί νέοι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη χώρα τους ή την πόλη τους για να βρουν δουλειά. Σίγουρα αυτό δεν είναι η ιδανική ευκταία κατάσταση, αλλά θα πρέπει να εφαρμόσουμε τα κατάλληλα μέτρα για να έχουμε μια πιο ισορροπημένη κατάσταση όσον αφορά την κινητικότητα αυτή των νέων και για να βοηθήσουμε τελικά του νέου να βρουν όντω μια πραγματική θέση εργασία. Αναφέρομαι πιο συγκεκριμένα στα άτομα εκείνα τα οποία εγκαταλείπουν πολύ γρήγορα το εκπαιδευτικό σύστημα, δεν συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα κατάρτισης και δεν έχουν εργασία. 15% είναι οι νέοι αυτοί στην Ευρώπη και καταλαβαίνω ότι ε, οι άνθρωποι αυτοί κινδυνεύουν πολύ περισσότερο από τους άλλους να αποκλειστούν κοινωνικά. Στην ίδια κατηγορία ανοίγουν, ανήκουν και οι μητέρες οι οποίες μεγαλώνουν μόνες τα παιδιά τους, καθώς επίσης και οι ανάπηροι. Μία άλλη σημαντική πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι το ότι, δεν υπά... το ότι υπάρχει μια αναντιστοιχία οτι δεν υπαρχει μια αναντιστοιχια αναμεσα στα εκπαιδευτικά συστήματα και τις πραγματικές ανάγκες αγοράς εργασίας. Θα πρέπει να γίνουν βιώσιμε μεταρρυθμίσει στην πολιτική εκπαίδευση. Η εκπαίδευση θα πρέπει να αποτελεί ένα πολύ σημαντικό μέσο για να γίνουν απαραίτητε επενδύσει για το μέλλον. Θα πρέπει να προσαρμόσουμε τα πανεπιστημιακά προγράμματα και τα προγράμματα των σχολείων για να αντιστοιχούν περισσότερο στι ανάγκε τη αγορά-εργασία. Για να επιτευχθεί όμω ο στόχο αυτό, θα πρέπει να παρέχονται καλύτερες υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και ήδη ο επαγγελματικό προσανατολισμό θα πρέπει να ξεκινάει από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και θα πρέπει να βασίζεται στα στατιστικά δεδομένα τη αγορά εργασία, δεδομένου του ποσοστού ενεργεία που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Και για να αντιμετωπίσουμε τη μάστιγα αυτή, νομίζω ότι θα πρέπει να πείσουμε περισσότερο τα κράτη-μέλη ότι οι επενδύσεις που κάνουν στους νέους δεν είναι χαμένα χρήματα, αλλά είναι μια πραγματική επένδυση για το μέλλον θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ένα υψηλό επίπεδο επαγγελματική κατάρτιση και πρακτική άσκηση για του νέου πτυχίουχου. Θα πρέπει να στηρίξουμε τι επιχειρήσει εκείνε που υποδέχονται στου κόλπου του νέου πτυχίουχου και θα πρέπει να προωθήσουμε περισσότερο τα συστήματα εκείνα τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν ποιοτικά προγράμματα πρακτική άσκηση βασιζόμενοι στα παραδείγματα της δικής μου χώρας, νομίζω ότι θα πρέπει να προωθήσουμε πολύ περισσότερο την πρακτική αυτή άσκηση για τους νέους πτυχίουχους και θα πρέπει να πείσουμε τους εργοδότες ότι πραγματικά έχουν συμφέρον να παρέχουν την πρακτική αυτή άσκηση στους πτυχίουχους. Κατά αυτόν τον τρόπο οι επιχειρήσεις μπορούν να αποκτήσουν στη συνέχεια έναν εργαζόμενο ο οποίος θα είναι καλά καταρτισμένος ο οποίος θα έχει τα απαραίτητα προσόντα για το πόστο το οποίο πρόκειται να καλύψει. Λοιπόν, να προωθήσουμε περισσότερο την όλη ιδέα της πρακτικής ε, άσκησης. Οι εργοδότες επίσης θα πρέπει να αναγνωρίσουν όλες αυτές τις δεξιότητες της άτυπης ανεπίσημης ε, μάθησης, δεξιότητες δηλαδή που κερδίσει κανείς εκτός επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος. Ό,τι κάνουν όλα τα κράτη-μέλη στον τομέα αυτό θα πρέπει να αξιολογηθούν. Θα πρέπει να γίνεται αυτό με μια συστηματική παρακολούθηση και όλοι οι πόροι που δαπανώνται θα πρέπει να ελέγχονται επίση πολύ προσεκτικά για να έχουμε αποτελεσματικά μέτρα παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να βοηθήσουν τους νέους προκειμένου να καταφέρουν να προσαρμοστούν περισσότερο στις ανάγκες εργασία μέσω ενό συστήματος πρακτικής άσκησης με τη συμμετοχή των επιχειρήσεων θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα θετικό επικοδομητικό πνεύμα προκειμένου να απτυχθούν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες όπως το ξέρουμε άλλωστε είναι αυτές οι οποίες δημιουργούν τις περισσότερες θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αυτές λοιπόν οι οποίες μπορούν να παρέχουν θέσεις απασχόληση στην νεολαία μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, ελπίζω ότι όλοι μας εδώ στην Επιτροπή Απασχόληση θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε ένα κείμενο το οποίο θα δώσει μια θετική όθηση, θα μας βοηθήσει να επιλύσουμε το πρόβλημα της ενεργείας των νέων και ελπίζω θα καταφέρουμε να προτείνουμε λύσεις οι οποίες θα είναι ελπιδοφόρες για τους νέους. Είμαι ανοιχτή στη μέση διαθεσή σας για ερωτήσεις παρατηρήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Στάιρουκ, αλλά προηγουμένως θα ήθελα να πω το εξής. Τώρα έτυχε να πέσει εσάς ο κλήρος στη δική σας έκθεση, κυρία Σεζερέσκα. Παρακαλώ μην το λάβετε αυτό ως προσωπική παρατήρηση, αλλά οι εκθέσεις αυτές είναι εκθέσεις πρωτοβουλίας, τις οποίες διαπραγματευόμαστε μεταξύ συντονιστών βάσει των ετοιμάτων των διαφόρων πολιτικών ομάδων και όπου προσπαθούν όλοι να είναι φιλικοί ε, για να αισθάνεται ο καθένας άνετα και να αναλαμβάνει τα θέματα που τον ενδιαφέρουν. Ταυτόχρονα όμως γνωρίζετε ότι εδώ στο Κοινοβούλιο και δικαίως υπάρχει μια ανησυχία γιατί πολλαπλησιάζονται εκθέσεις πρωτοβουλίας που δεν έχουν σχέση με άμεση νομοθετική δραστηριότητα. Δηλαδή, μια έκθεση νομοθετικής πρωτοβουλίας τι σκοπό έχει. Είτε να προλιάνει το έδαφος είτε να προετοιμάσει μια ε, πρωτοβούλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είτε να αντιδράσει σε ένα κείμενο που έχει βγάλει για διαβούλευση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ δεν συμβαίνει τίποτα από όλα αυτά. Για λόγους χρονοδιαγραμμάτος. Ε, καλός ή κακός, επειδή τα πράγματα είναι σοβαρά, ε, έχουν επιταχυνθεί οι διαδικασίες. Και επίσης και εν ώψη των ε, αποφάσεων, μάλλον μετά τις αποφάσεις 7 και 8 Φεβρουαρίου του Συμβουλίου και η συγκήτρια δείχνει ότι έχει πλήρη επίγνωση αυτής της κατάστασης ε, και των εξελίξεων. Λοιπόν, αυτό το τραβηχτικό δικαίωμα λοιπόν που έχουμε εμείς πλέον και ξεκίνησε με την έκθεση πρωτοβουλίας θα πρέπει να το αξιοποιήσουμε όσο γίνεται περισσότερο. Τι εννοώ. Εσείς και οι και μαζί με την εισηγήτρια σε αυτό το κύκλο συζητάτε να δούμε ποιο είναι το συγκεκριμένο μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε στο συνολικό και παγκόσμιο πλαίσιο που ζούμε τώρα και στις όλες τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται εμείς, τι μήνυμα θέλουμε να στείλουμε για να δείξουμε ότι είμαστε χρήσιμοι. Διότι δεν είμαστε δημοσιογράφοι, Ε, θα πρέπει να έχουμε χρήσιμες αναλύσεις βέβαια. Καλές είναι οι διαπιστώσεις και οι αναλύσεις, αλλά εμείς δεν είμαστε σχολιαστές. Είμαστε πολιτικοί, ηθήνοντες. Και αν θέλουμε να αξιοποιήσουμε το έργο της συναδέλφου συγγήτριας, θα πρέπει να καταλήξουμε, να έχουμε κατασταλαγμένα 4-5 πολύ συγκεκριμένα μηνύματα, να στείλουμε ως Επιτροπή Απασχόλησης, πέραν των όσων ήδη είναι επιτάπητος. Θα δώσω λόγο στη Γιούτα Στάιροκ, μετά στην Άδεια Χίρς. Άλλος κανείς. Αυτή προς το παρόν. Η ε, Γιούτα, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και για το σχόλιο σας και τις υποδείξεις. Η κυρία Ρέγνερ είναι σκιώδη συγγήτρια δική μας και δυστυχώς κολλείεται σήμερα παρευρεθεί. Λυπάται πάρα πολύ γι' αυτό και με παρακάλεσε να παρουσιάσω τις θέσεις της. Ε, θέλει να ευχαριστήσει την εισηγήτρια για την εργασία της για αυτό το τόσο πολύ σημαντικό θέμα. Ξέρει ότι υπήρξε και χρονική πίεση η κυρία Ρέγνερ ως σκιώδη ηγήτρια όμως θα ήθελε να είχε συμπεριληφθεί πολύ περισσότερο και πολύ νωρίτερα σε αυτή την προσπάθεια. Το σχέδιο της ηγήτριας αγαπητοί συνάδελφοι είναι καλό σε γενικές γραμμές και καλό είναι να έχουμε μια συνολική θεώρηση και προσέγγιση για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της ανεργίας των νέων. Γιατί είναι πολλές οι αιτίε και ποικίλε ε, και πολλές οι ανάγκες των νέων και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Όλα αυτά λοιπόν Λαμβάνονται υπόψη στην έκθεση και η συμμετοχή όλων των ενεχομένων είναι απαραίτητη και αποφασιστική. Η Εύελιν Ρέγνερ είναι πολύ επικριτική απέναντι σε ιδιωτικές εταιρείες εξέφρασης εργασίας, γιατί αυτό είναι ενισχυτική εξέλιξη. Και οι νέοι μας, όσο και οι υπόλοιποι, χρειάζονται ε, δουλειά υψηλής ποιότητας με αντίστοιχες αμοιβέ. Γι' αυτό υπάρχουν οι ε, κρατικοί οργανισμοί ε, απασχόλησης. Επανειλημμένα ε, μιλάει η συγγήτρια για ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των νέων. Εντάξει, ποιος θα διαφωνήσει σε αυτό, αλλά υπάρχει το θέμα της μαζικής ανεργίας, το οποίο δεν λύνεται με αυταπασχόληση είναι σχετικά μικρό το ποσοστό των νέων που αμέσως μετά ε, το τέλος της εκπαίδευσης τους θέλουν να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση και έχουν και τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να το κάνουν. Ήδη από τώρα υπάρχει και ένα ε, φαινόμενο των εικονικών αυτοαπασχολουμένων ε, που είναι μια στρεβλή εξέλιξη στην αγορά εργασίας και γι' αυτό φταίνε συχνά οι εργοδότες. Το ξέρω ότι δεν είναι πρόθεση της εισηγήτριας ε, να το δικαιολογήσει αυτό, αλλά θα πρέπει να πούμε ότι οι νέοι θα πρέπει να ε, απασχολούνται σε θέσεις εργασίας αξιοπρεπής και με σωστή αμοιβή. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το τρίγωνο που ονομάζεται Πανεπιστήμια Εργοδότες ε, και νέοι Ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση οικονομική. Πολλές επιχειρήσεις ε, περνούν κρίση, αλλά θα πρέπει να αναλάβουν και εταιρείε τι ευθύνε τους για να ε, εκπαιδεύονται σωστά οι εργαζόμενοι και να ε, φτάνουν στην αγορά εργασίας. Η κυρία Ρέγνερ θα κάνει και τροπολογίε και προσβλέπει συνεργασία με τις άλλες πολιτικέ ομάδε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Όντω η κυρία Ρέγνερ με είχε παρακαλέσει να αλλάξουμε τη σειρά συζήτηση στην ημερήσια διάταξη αυτού του θέματος για να είναι παρούσα. Αλλά, ειλικρινά, θα ήθελα ως κανόνα να προσανατολιζόμαστε στα αιτήματα των εισηγητών όταν πρόκειται να αλλάξουμε τη σειρά. Αν μπούμε τώρα και ε, σε αυτό τον κύκλο του, του να αλλάζουμε με βάση τα αιτήματα και τις επιθυμίες των σκιωδών ε, εισηγητών, τότε θα πρέπει να τετραγωνίσουμε τον κύκλο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι άδεια Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ την εισηγήτρια για την έκθεσή της. Πάντα είναι δύσκολο το έργο να κάνει κανείς μια έκθεση που να καλύπτει τα πάντα για ένα θέμα το οποίο εξελίσσεται τόσο γρήγορα. Εμείς γράφουμε εκθέσεις και εκθέσεις πρωτοβουλίας για τον έξω κόσμο, όχι να τις διαβάζουμε μεταξύ μας. Και όποιος διαβάζει για πρώτη φορά αυτό το θέμα, ε, ως πολίτης, ε, για να δει τι σημαίνει ενεργεία των νέων, με την παρούσα έκθεση έχει μια πολύ καλή εικόνα. Κάτι άλλο που θυμάμαι εγώ από την έκθεση που είχα κάνει για τη μετανάστευση. Βεβαίω θα πρέπει να βάζουμε και κάποια κέντρα βάρους και να εστιάζουμε γενικά η έκθεση αναφέρει όλα τα προβλήματα. Τώρα, στη συζήτηση με τους σκιώδεις εισηγητές, θα δούμε ποια είναι εκείνα τα θέματα που θέλουμε να επιμείνουμε περισσότερο. Ότι αυτό είναι το βασικό μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε προς τα έξω, προς την Κομισιόν, το Συμβούλιο κλπ. και με τις συμβαστικές τροπολογίες. Πάντως θα τα καταφέρουμε. Είμαι πεπισμένη. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για την κινητικότητα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την άποψή μου, αυτό λίγο χάνεται στη συνολική συζήτηση. Υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Έχουμε θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν καλύπτονται. Ψάχνουμε νέους με προσόντα, με δεξιότητες. Θα πρέπει να το πούμε και αυτό να συναντήσουν οι προσφορές τη ζήτηση. Και το Κοινοβούλιο μπορούμε να προσθέσουμε ιδέες πέρα από τα καλά κατά τα άλλα προγράμματα που έχουν τα κράτη-μέλη. Μπορούμε και εμείς να βάλουμε το λιθαράκι μας. Κάτι που μου αρέσει πολύ στην έκθεση είναι η διάκριση που γίνεται. Για ποιο λόγο είναι οι νέοι άνεργοι, όχι επειδή είναι νέοι και μόνο. Εντάξει, το ένα είναι αυτό δεν έχουν οι νέοι συχνά εκπαίδευση, κατάρτιση, αποχωρούν νωρί από το σχολείο. Αυτά είναι τελείως διαφορετικά μέτρα που χρειάζονται. Αλλά υπάρχουν και νέοι που είναι πτυχιούχοι και παρόλα αυτά άνεργοι. Οπότε εκεί μπαίνει η κινητικότητα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το θέμα της αυταπασχόλησης, πολύ καλό. Υπάρχουν καλές ιδέες και εδώ και ιδιαίτερα στον τομέα των μέσων ενημέρωσης και το διαδίκτυο, πολλοί είναι οι νέοι που δραστηριοποιούνται και απασχολούνται με εταιρείε δικές τους. Καλό είναι να το αναφέρουμε και αυτό. Πολύ ωραίο. Και ένα τελευταίο. Επίσης καταφέραμε πάρα πολύ καλά να πούμε ότι θα πρέπει να συμμετέχουν όλοι, σχολεία, πανεπιστήμια, εργοδότες, συνδικάτα, κοινωνικοί εταίροι, ε, γραφεία ευρέσεως εργασίας. Βεβαίω, ο εκάστοτε ο ΑΕΔ, α πούμε, αλλά ξέρουμε πολύ συχνά πόσο μεγάλο είναι ο φόρτο. Ε, γιατί όχι. Και βεβαίω θα πρέπει να υπάρχουν και ιδιωτικά γραφεία ευρέσεω εργασία, Αφήστε που ε, πολλές φορές είναι και ποιοτικότερα των κρατικών. Δεν μπορούμε να πούμε από την ε, αρχή από χέρι ότι αποκλείουμε ε, τα ιδιωτικά κέντρα. Δεν θέλουμε παροπίδες εδώ. Ο κόσμος ψάχνει δουλειά. Άμα μπορεί κάποιος να του βρει δουλειά, έστω και ιδιώτης, τι πειράζει θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα ο νέος να μπει ε, σε ένα επάγγελμα, να μπει στην αγορά εργασίας. Αυτό χρειαζόμαστε και όχι παροπίδες. Μέχρι τώρα δεν το έχουμε καταφέρει αυτό. Πρέπει να βρούμε ένα νέο τρόπο. Ευχαριστώ πολύ και χαίρομαι για τη συνεργασία που θα έχουμε στη συνέχεια. Υπάρχουν άλλοι που θέλουν το λόγο. Δεν βλέπω κανέναν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να πάρει το λόγο. Σας καλύψαμε. Θα μιλήσετε, ναι, όχι. Λοιπόν, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και σας ευχαριστώ που δίνετε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εν γέννη εξ ονόματος Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορώ να σας πω ότι συμφωνούμε με το περιεχόμενο της έκθεσης. Ωστόσο, εν συντομία, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα από τα ζητήματα στα οποίο αναφέρθηκε η συγγήτρια όσον αφορά την χρησιμότητα κάποιων τεχνητών συστημάτων. Νομίζω ότι θα πρέπει να θεωρήσουμε τα μέτρα αυτά ως συμπληρωματικά προς τα υπόλοιπα μέτρα τα οποία έχουν ως στόχο να τονώσουν την οικονομία. Δεν νομίζω λοιπόν ότι η εγγύηση για την νεολαία θα πρέπει να θεωρηθεί ως τεχνητό μέσο, αλλά συμπληρωματικό μέσο. Πέρα από αυτό, θα ήθελα σύντομα να σας ενημερώσω για το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την εφαρμογή του πακέτου για την απασχόληση των νέων όπου έχουμε μια πρόταση σύσταση του Συμβουλίου για την εγγύηση για την νεολαία, μια πρόταση για διαβούλευση των κοινωνικών εταίρων για ποιοτικά εκπαιδευτικά προγράμματα, ποιοτικά μάλλον προγράμματα πρακτικής άσκησης, Επίσης, τη δημιουργία μιας συμμαχίας για προγράμματα μαθητείας και το καθεξής. Όσον αφορά την εγγύηση για την νεολαία, έχουμε μια, έχουμε μια σύσταση του Συμβουλίου, η οποία έχει εγκριθεί, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι έχουμε ε, μια υποστήριξη υψηλού επίπεδου και από τα κράτη-μέλη. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται τώρα την ανάλυση κάποιων προτάσεων πρόσκληση υποβολής προτάσεων, δηλαδή στα πλαίσια της εγγύησης για την νεολαία. Έχουμε λάβει 140 αιτήσει αυτή τη στιγμή, 15 εκ των οποίων θα επιλεγούν στη συνέχεια τις επόμενες εβδομάδες και περιμένουμε ότι ε, τα πρώτα σχέδια θα μπορούν ήδη από το Σεπτέμβριο του 2013 να αρχίσουν να εφαρμόζονται. Και είμαστε πεπισμένοι ότι η εμπειρία που θα αποκομίσουμε από τα πιλωτικά αυτά προγράμματα θα βοηθήσει πολύ τα κράτη-μέλη και ιδίω την τοπική αυτοδιοίκηση στο να δημιουργήσει προγράμματα εγγύησης για την νεολαία σε ευρύτερη κλίμακα, σε μεγαλύτερη κλίμακα. Όσον αφορά τώρα την πρακτική άσκηση. Ολοκληρώθηκαν οι διαβουλεύσεις το Φεβρουάριο, οι κοινωνικοί εταίροι είχαν τη δυνατότητα να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για ένα ποιοτικό πλαίσιο, αλλά τελικά αποφάσισαν να μην κάνουν κάτι τέτοιο, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τώρα την δυνατότητα να παρουσιάσει τη δική της την πρωτοβουλία και αυτό ακριβώς θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάνουμε μια αξιολόγηση αντικτύπου αυτή τη στιγμή και θα κάνουμε και μια τελική πρόταση στα τέλη του έτους όσον αφορά την πρακτική άσκηση. Τώρα για την συμμαχία για τα προγράμματα μαθητείας. Βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες και η συμμαχία αυτή θα αρχίσει να λειτουργεί από τις αρχές Ιουλίου, από την 3η Ιουλίου. Την 3η Ιουλίου έχουμε στο, στην Λειψία της Γερμανίας μια συνεδρίαση υψηλού επίπεδου σχετικά με τη συμμαχία αυτή για τα προγράμματα μαθητείας. Και έπειτα έχουμε και ένα άλλο πρόγραμμα εξυγχρονισμού του συστήματος EURES με στόχο να βελτιώσουμε την κινητικότητα των νέων και αναφερόμαστε εκεί και στην κινητικότητα των νέων που συμμετέχουν σε προγράμματα μαθητείας και πρακτικής άσκησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται αυτή τη στιγμή διαφόρους τρόπους προκειμένου να περιλάβει και αυτά τα προγράμματα στα προγράμματα κινητικότητα. Ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο έχει πάλι η συγγήτρια. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα απαντήσω πρώτα στην Κομισιόν. Μήπως δεν κατάλαβα καλά ή μήπως δεν ήταν ακριβής η διερμηνία. Εγώ δεν είπα ότι η εγγύηση για την νεολαία είναι τεχνητό λέει πρόγραμμα το οποίο δεν το χρειαζόμαστε. Εγώ υποστηρίζω αυτή την πρωτοβουλία αλλά σας τονίζω ότι πρόκειται για ad hoc λύση γιατί τα 6 δισεκατομμύρια που προβλέπονται για την, α, ε, το εκατομμύριο προβλέ, τα 6 δισεκατομμύρια προβλέπονται αν τα χωρίσουμε σε όλους τους νέους άνεργους θα έχει ο καθένας πολύ χαμηλό ποσό Μπορούμε με το ποσό αυτό λοιπόν να αλλάξουμε την κατάσταση αυτών των νέων στην αγορά εργασίας. Δεν νομίζω. Νομίζω λοιπόν ότι πρόκειται για λύση που δεν λύνει τίποτα. Τώρα θα αναφερθώ σε αυτά που είπαν οι συνάδελφοι, τα μέλη της Επιτροπής μας δηλαδή. Καταρχάς ευχαριστώ όλους εκείνους που έλαβαν το λόγο, την κυρία Στέινρουκ, ελπίζω να προφέρω καλά το όνομά της, αλλιώς ζητώ συγγνώμη. Εσείς τονίσατε ιδιαίτερα τις ε, εθνικές δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες ευρέσεως εργασίας. Εδώ όμως Υπάρχουν πολιτιστικές διαφορές. Στη δική μου χώρα, παραδείγματος χάρη, δουλεύουν πολύ καλά οι υπηρεσίες αυτές και οι νέοι εποφελούνται από τις υπηρεσίες αυτές. Αλλά εγώ θα ήθελα μια λύση που να τους ικανοποιεί όλους. Και απ' την άλλη υποστηρίζω ότι οι νέοι πρέπει να έχουν δικαίωμα επιλογής μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής υπηρεσίας ευρέσεως εργασίας. Κυρία Χίρς, αναφερθήκατε στην κινητικότητα μέσα στην Ευρώπη. Για μένα είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, ούτε αυτό είναι η ιδεώδης λύση. Ούτε και τίποτα πολύ εύκολο, γιατί οι νέοι για να μετακινηθούν καμιά φορά πρέπει να μετακινήσουν και τις οικογένειές τους. Δεν είναι λοιπόν ούτε αυτό η ιδεώδης λύση, ελπίζω όμως ότι θα μπορέσουμε να το ξανασκεφτούμε και να βρούμε κάποια συμβιβαστική λύση αποδεκτή επαναλαμβάνω για όλους. Τέλος, για αυτά που είπε η κυρία Πρόεδρος. Δεν συμφωνώ πάντοτε με την Πρόεδρο, αλλά σας διαβεβαιώνω ότι δεν, παρερμη, δεν ερμήνευσα αυτά που είπατε για μένα όσο αυτά που είπατε όσο κάτι που ψέγατε σε μένα. Ξέρω ότι πολλά μέλη της Επιτροπής Απασχόλησης έχουν ασχοληθεί με το θέμα και βλέπουμε ότι η κατάσταση αντί να βελτιώνεται χειροτέρεψε. Συμφωνώ λοιπόν με την θέση ότι οι εκθέσεις πρωτοβουλίας που είναι περιορισμένες και ως προς το μήκος τους οι εκθέσεις λοιπόν πρωτοβουλίας συμφωνώ ότι δεν μας επιτρέπουν να εκφράσουμε αυτά που θέλουμε ελεύθερα. Ευχαριστούμε. Βιωρία κατάθεση τροπολογιών λίγη στις 22 Μαΐου στις 2 το απόγευμα. Θα εξεταστούν οι τροπολογίες στις 20 και 21 Ιουνίου οι συμβιβαστικές τον Ιούλιο, αρχές Ιουλίου και ολομέλεια τον Σεπτέμβριο. Τελειώσαμε και με αυτό το σημείο τώρα και πάμε στο επόμενο και βασικότατο γνωμοδότηση του συναδέλφου Χρίστενσεν προς την Επιτροπή Πολιτισμού για την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για την νεολαία 2010-2012. Στην Επιτροπή Πολιτιστικών ο εισηγητής επί της ουσίας είναι, είναι πώς να το πω, ποιος είναι. Δεν ξέρω. Θα σας το πω μετά. Λοιπόν, ο κύριος Χρίστενσεν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι προφανές ότι αντιμετωπίζουμε τεράστιες προκλήσεις. Η ανεργία των νέων στην Ευρώπη έχει διπλασιαστεί. τα τελευταία χρόνια. Χρειάζεται λοιπόν κάποια στρατηγική. Η Κομισιόν πρότεινε μια τέτοια στρατηγική για ενδυνάμωση, ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών μελών για τους νέους 2010-2012. Θέλουμε να δώσουμε στους νέους περισσότερες ευκαιρίες για πρόσβαση στην ε, αγορά εργασίας. Ε, να ενθα, τους ενθαρρύνουμε να συμμετάσχουν πιο ενεργά. Αρχικά προβλέπαμε την περίοδο 2010-2018 με πρώτο κύκλο 10 με 12 που εξετάζουμε εδώ. Πρέπει να κάνουμε λοιπόν την αποτίμηση αυτού του πρώτου κύκλου και να δούμε τι προβλέπουμε για τον επόμενο τριετή κύκλο. Για το ίδιο πάντα θέμα την νεολαία. Η γνωμοδότησή μου απευθύνεται λοιπόν στην Επιτροπή Πολιτιστικών, αλλά δυστυχώς δεν συνεργαστήκαμε επαρκώς με την Επιτροπή αυτή, ενώ το θέμα της αγοράς εργασίας είναι ουσιώδες. ουσιώδες. Γιατί τέθηκαν προβλήματα δικαιοδοσιών και δεν καταλήξαμε σε καμία ικανοποιητική μεθοδολογία. Ξέρετε ότι όταν γράφονται τέτοιου είδους χρωμοδοτήσεις έχουμε πολλούς περιορισμούς και γι' αυτό χρειάστηκε να περιοριστώ στα αυστηρά απαραίτητα. Λοιπόν, η στρατηγική για την νεολαία πρέπει να δίνει στους νέους πιο ισότιμες ευκαιρίες πρόσβασης στην ε, αγορά εργασίας και στην κοινωνική προστασία. Με στόχο βέβαια κάποιο απτό αποτέλεσμα. Η στρατηγική λοιπόν αυτή με την τωρινή κρίση έγινε ακόμα πιο σημαντική και την ψηλή ανεργία. Ελπίζω να μπορέσουμε να γεφυρώσουμε τον προηγούμενο τριετή κύκλο με τον επόμενο έτσι ώστε η στρατηγική για την νεολαία να, αποτε... να από μια νέα όθηση. στην γνωμοδότησή μου βλέπουμε τα πράγματα λίγο πιο μακροπρόθεσμα και χαίρομαι ιδιαίτερα για τη συνεργασία που είχαμε τους Κιώδης. Ευχαριστώ. Η κυρία ε, Βερόνικα Λόπε Φοντανιέ και μετά θέλει κανείς άλλο το λόγο. Η κυρία Χίρς ε, ε, που θα μας γίνει ειδική για τους νέους στο τέλος. Η κυρία Βερόνικα Ρόπε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κλείνει το μικρόφωνο της η ομιλήτρια. Συμφωνώ με τον εισηγητή ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν κανείς καταρτίζει μια γνωμοδότηση να επεκτείνεται γιατί είναι πάρα πολύ περιορισμένες οι δυνατότητες που έχουμε από πλευράς έκτασης της γνωμοδότησης ιδιαίτερα για τους νέους και την ανεργία των νέων γιατί αυτό το κομμάτι μας αναλογεί μας ως Επιτροπή Απασχόλησης. Σήμερα η στρατηγική για την νεολαία ε, περιέχει κάποια στοιχεία απασχόλησης που είναι πάρα πολύ απαραίτητα. Ανισχυτική είναι η αύξηση της ανεργίας των νέων και σε κάποιες χώρες και δυστυχώς μεταξύ αυτών είναι και η δική μου το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι φλέγον και προτεραιότητα. Μια στρατηγική λοιπόν για τους νέους είναι πάρα πολύ σημαντική αλλά επίσης θα πρέπει να μελετήσουμε την κατάσταση της ανεργίας, πώς εξελίσσεται και πώς αντιμετωπίζεται. Όπως είπε και ο εισηγητής, θα πρέπει να βρούμε με ποιο τρόπο θα συμμετέχουν περισσότερο οι νέοι μας στην κοινωνία. Στην Αραγωνία, από όπου κατάγομαι, έχουμε επίσης πολύ μεγάλη ανεργία των νέων. Ίσως από τα χαμηλότερα ποσοστά στην Ισπανία, αλλά είναι διπλάσια η ενέργεια των νέων σε σχέση με τους μεγαλύτερους. Και μόλις βγήκε μια έρευνα που πρέπει να μας κάνει να σκεφτούμε. Τι λέγει αυτή, ότι περίπου οι μισοί νέοι από την Αραγωνία, και αυτό μπορεί να μεταφερθεί και στην υπόλοιπη Ισπανία, έχουν απευδίσει πλέον, δεν ψάχνουν καν για δουλειά οι μισοί. Θεωρούν ότι σιγά μη βρω δουλειά ποτέ, οπότε δεν ψάχνω κιόλα. Ε, βεβαίως είναι γεγονός ότι Μερικοί έχουν επιστρέψει στην εκπαίδευση ή ε, συνεχίζουν τις σπουδές τους σε περίπτωση που τις είχαν ε, διακόψει. Γι' αυτό αυτή τη στιγμή στην Ισπανία έχει μειωθεί η αποχώρηση από το σχολείο. Για ποιο λόγο, ακριβώς επειδή δεν υπάρχει δουλειά παραμένουν στο σχολείο. Ε, παλαιότερα βρίσκανε δουλειά και φεύγανε νωρίτερα από το σχολείο. Άλλοι μετανάστευσαν. Πρέπει όμως να βρούμε κάθε φορά την κατάλληλη λύση. Καλό είναι και θετικό να εκπαιδεύονται οι νέοι μας και να μορφώνονται, αλλά κάπου ε, όλα αυτά να αξιοποιούνται, να προσαρμόζονται σε μια ε, δουλειά, θέση εργασία στη συνέχεια. Συνεπώς, καλό είναι που υπάρχει μια τέτοια στρατηγική και η Επιτροπή μας θα πρέπει να πει πολλά για τους νέους. Αυτά και τελείως. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ήρς έχει το λόγο και ο Τόμας Χέντελ στη συνέχεια. ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς ευχαριστώ πολύ και τον εισηγητή μας για τη γνωμοδότησή του. Με ενδιαφέρον τη διάβασα. Και βέβαια αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλές επικαλύψεις με την έκθεση. Παρ' όλα αυτά εμείς ως Επιτροπή ε, απασχόλησης θα πρέπει να γνωμοδοτήσουμε στην Επιτροπή Πολιτιστικών Υποθέσεων ακριβώς ε, εστιάζοντας στην απασχόληση. Εντάξει, το ξέρω ότι υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα που παίζουν ρόλο στη στρατηγική για την νεολαία, διότι οι νέοι δεν υπάρχουν μόνο για να μορφώνονται έτσι ώστε να μπορούν να δουλέψουν. Έχουν και άλλες δραστηριότητες στη ζωή τους, μέχρι και πολιτική στράτευση. Ε, αλλά εμείς ως Επιτροπή Απασχόλησης πρέπει να εστιάσουμε σε αυτό ε, το θέμα της εργασίας. Νομίζω έχουν υποθεί τα περισσότερα, τα σημαντικότερα και με ένα τέτοιο χρονικό ορίζοντα και κοιτάμε και άλλα προβλήματα. Εντάξει, η εγκατάλειψη του σχολείου ε, είναι ένα θέμα που θα παραμείνει, δεν εξαφανίζεται. Στο σημείο 5 αναφέρεστε στην πρακτική άσκηση. Ε, το θέμα είναι τώρα τι εννοείται ποιοτικό πλαίσιο η πρακτική άσκηση έχει ένα χαρακτήρα μετακπαίδευση. Είναι ε, μια περίοδος όπου κάποιος συγκεντρώνει γνώσεις. Όταν είναι ένας ασκούμενος, δεν σημαίνει ότι βγάζει φωτοτυπίες όλη μέρα ή φτιάχνει καφέδες, γιατί υπάρχει και αυτό. Το έχουμε ξανασυζητήσει. Και άσκηση θα πρέπει πάντα να είναι αμοιβόμενη, όχι άμυστη γιατί υπάρχουν και διεθνείς οργανισμοί που δεν έχουν χρήματα για να πληρώνουν με σωστό τρόπο και αξιοπρεπή όλους τους νέους που θέλουν να κάνουν άσκηση σε αυτούς τους οργανισμούς. Βεβαίως και να αμείβεται, ιδιαίτερα όταν διαρκεί ε, περισσότερο από τρεις μήνες περίπου, θα, πρέπει να είναι άμυστη αυτή η περίοδος. Αν θέλει κάποιο να έρθει ένα τρίμηνο για να πάρει μια γεύση του τι είναι αυτή η δουλειά, δεν θα πρέπει να τον αποτρέπουμε, αλλά αν είναι μεγαλύτερη διάρκεια πρέπει να αμείβεται η άσκηση αυτή. Αυτή τη στιγμή κάποιο παρέχει ε, υπηρεσίες. Είπαμε μετά το τρίμηνο να πληρώνεται. Αν σε λιγότερο από τρει μήνες κάποιο θέλει απλώς να κοιτάξει πώς είναι αυτή η δουλειά για να αποφασίσει, ε, προσοχή να μην καταστρέψουμε και θέσει εργασία έτσι και διαδρομίε. Αυτά όλα τα άλλα πολύ ωραία, πολύ σημαντικά και συμφωνούμε σε μεγάλο βαθμό και με την έκθεση για την ενεργεία των νέων επικαλύπτονται πολύ. Ευχαριστώ ο Τόμας Έντελ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όλε Κρίστενσεν με την έκθεση αυτή έχει ένα περιορισμό σε χαρακτήρες και σε μέγεθος της ε, γνωμοδότησης. Έχει καλύψει τα βασικότερα θέματα. Για τα περαιτέρω μπορούμε να τον βοηθήσουμε με τροπολογίες για να μπορέσει να τα εντάξει στην έκθεσή του, αν πρέπει επιγόντως να μπουν. Ιδιαίτερα σημαντικό ε, είναι το γεγονός ότι εστιάζει σε ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού Βλέπουμε στην Ευρώπη διάφορους κυνηγού κεφαλών που τρέχουν και βρίσκουν τα καλύτερα μυαλά και τα φέρνουν ε, στα κέντρα στην Ευρώπη και απομένουν εκείνοι που κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό ή με χαμηλή μόρφωση ε, κτλ. τα Αυτό κατά την άποψή μας έχει τον κίνδυνο της διαρροής εγκεφάλων, το brain drain και αυτό θα πρέπει να το πούμε και στην Επιτροπή Πολιτισμού και να το επισημάνουμε. Το δεύτερο αφορά αυτό που ανέφερε προηγουμένως η κυρία Χίρς. Εγώ το βλέπω από διαφορετική σκοπιά, κυρία Χίρς και αγαπητοί συνάδελφοι. Στο θέμα του ποιοτικού πλαισίου για την πρακτική άσκηση θα πρέπει να δούμε να μην εκφυλιστεί αυτή η κατάσταση και να μην χρησιμοποιούνται οι νέοι, να μην τους εκμεταλλεύονται ουσιαστικά σε ασκήσεις ε, πρακτικές που δεν μαθαίνουν τίποτα, δεν βγάζουν λεφτά και επίσης ε, ε, στη συνέχεια δεν αποκομίζουν κανένα προσόν που να μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν στη δουλειά τους. Τους ξέρουμε αυτούς από τα περασμένα χρόνια, τους απλήρωτους ασκούμενους και θα πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε κάποια κριτήρια για αυτό το θέμα, αλλιώς κινδυνεύουμε. Κατά τα άλλα συμφωνούμε. Συμφωνώ γενικά με την εισηγήτρια της προηγούμενης έκθεσης. Αυτά τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ είναι πάρα πολύ λίγα λεφτά. Δηλαδή, αν δούμε πόσοι είναι οι νέοι άνεργοι, αναλογούν 800 ευρώ στον καθένα. Ενώ η Ευρώπη για να έχει μια σωστή θέση μόρφωσης, ε, αυτό κοστίζει 15 με 20.000 ευρώ το χρόνο κατάτομο. Ακόμα και αν εξαντληθεί το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, δεν ξέρω αν θα καλυφθεί αυτό. Ιδιαίτερα σε χώρες ε, που ε, είναι υποχρεωμένοι σήμερα να εργάζονται με πάρα πολύ μεγάλους περιορισμούς στα οικονομικά τους και δεν μπορούν να συγχρηματοδοτήσουν. Ακόμα και αν ε, είναι σχετικά ευέλικτες οι ρυθμίσεις, κάπου πρέπει να το γράψουμε και αυτό στην έκθεση. Και ένα τελευταίο, για να βρεθεί λύση, θα πρέπει στο μέλλον να υπάρχει μια στρατηγική που να ασχολείται ε, και με τις επενδύσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Και αυτό είναι σημαντικό. Το έχουμε πει και σε προηγούμενες εκθέσεις, κυρίως ο Αλεχάνδρος Σέρκας και η συνάδελφος Μπερές. Ε, εδώ μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό και να δείξουμε ότι έχει συνέχεια η Επιτροπή μας στις εκθέσεις της. Τέλος, θεωρώ πολύ σημαντικό το θέμα της συμπερίληψης των κοινωνικών εταίρων σε αυτή την προσπάθεια είναι βασικοί παίκτες εδώ για να δίνουν ε, μια πραγματική προοπτική ε, του μέλλοντος στους νέους μας. Ευχαριστώ. Μήπως θέλει κανείς άλλος να λάβει το λόγο. Όχι. Η Κομισιόν. Η κυρία Κάλμαν. Λοιπόν, ε, δεν λέγομαι έτσι αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν. Συμφωνούμε με τα συμπεράσματά σας εδώ ότι η ανεργία των νέων είναι τεράστιο πρόβλημα και από αυτά που είπε ήδη και ο συνάδελφος από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης Βλέπετε ότι έχουμε ήδη αναλάβει ορισμένες πρωτοβουλίες στον τομέα της παιδείας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρέπει να συνδυάσουμε τις προσπάθειές μας και να συνεργαστούμε στον τομέα της παιδείας και για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Um, Και επίση είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι δεν θα αποκλείεται κανείς, δεν θα χάσουμε κανέναν. Όλα αυτά για να πούμε ότι η ανεργία είναι πολύ πολύ πλοκό πρόβλημα. Και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ό,τι εργαλεία διαθέτουμε για να την καταπολεμήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Χρίστενσεν. Ευχαριστώ και εγώ και τους σκιώδεις όλους για τα σχόλιά τους προς την εισηγησή μου. Συμφωνώ με την κυρία Φωντανή που μας είπε ότι υπάρχει το παράδειγμα της Αραγωνίας όπου πολλοί νέοι απελπίστηκαν πια. Αυτό είναι ο μεγάλος κίνδυνος. Αν δεν βρίσκουν πια λόγο να σηκωθούν το πρωί ή να πάνε στο σχολείο και το πανεπιστήμιο ή να πάνε σε κάποια δουλειά, τότε δεν γίνεται τίποτα. Πρέπει λοιπόν να επενδύσουμε σε αυτούς σε πολύ μεγάλο βαθμό τα 6 δισεκατομμύρια που προτείνει η Κομισιόν δεν είναι τίποτα βέβαια. Πρέπει να επενδύσουμε στο μέλλον. Αν δεν το κάνουμε και δεν επενδύσουμε σε αυτούς τους νέους, το πρόβλημα θα χειροτερέψει ακόμα περισσότερο στο μέλλον. Θα γίνουν οι νέοι αυτοί τελείως παθητικοί, θα μας λείπει το εργατικό δυναμικό και Γι' αυτό συμφωνώ ότι πρέπει να επενδύσουμε στους νέους. Επίσης συμφωνώ και με την κυρία Κίχ ότι ότι λέγω όταν μιλάμε για δωρεάν υπηρεσίες ή εργασία αυτό μπορεί να είναι ανησυχητικό, αν και θα μπορούσε να είναι και αυτό μια λογική πρόταση, αλλά γνωρίζουμε ότι πρέπει να αποφύγουμε τη δημιουργία νέου πρόσθετου στρώματος εκμετάλλευσης των νέων. Υπάρχουν, μπορεί να υπάρχουν μαθητείες απλήρωτες που να είναι θετικές, αλλά δεν πρέπει να είναι οι μόνες που θα προωθήσουμε. Ευχαριστώ τον Τόμας για όσα μας είπε. Συχνά μιλάμε για νέους με πολλά προσόντα, μορφωτικά προσόντα, αλλά μιλάμε και για νέους που εργάζονται χωρίς σχεδόν να πληρώνονται. Πρέπει τα κράτη-μέλη να επενδύσουν στο μέλλον αυτών των νέων. Αυτά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, <laughs> στην Επιτροπή Πολιτιστικών ο κύριος Παπα-Νικολάου είναι ο αρμόδιος επί της ουσίας και χθες ακούσαμε και την Επίτροπο κυρία Βασιλείου που μας ανέφερε τις πρωτοβουλίες της Κομισιόν και τη σχετική της δήλωση μέσα στα γενικότερα πλαίσια της στρατηγικής της Κομισιόν. Τώρα το χρονοδιάγραμμα. Διορία κατάσταση τροπολογιών λίγη στις 6 Μαΐου στις 2 το απόγευμα. Στις 12. Ε? Και ψηφοφορία στις 30 Μαΐου. Εδώ έχει ένα λάθος στα έγγραφα εδώ μπροστά μου. Λέει ότι θα ψηφίσουμε Απνό είναι απλή γνωμοδότηση, αλλά τέλος πάντων. Τα υπόλοιπα είναι όπως σας είπα. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα στην ώρα της ψηφοφορίας ακριβώς όπως προβλεπόταν και με δύο λεπτά νωρίτερα μας, δύο λεπτά νωρίτερα. Θέλετε να κάνουμε διάλειμμα δύο λεπτών ή όχι. Να περιμένουμε. Διάλειμμα δύο λεπτών. Μάλιστα, αγαπητοί συνάδελφοι, εφόσον είστε τώρα όλοι στην αίθουσα, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Να λοιπόν, ξεκινήσουμε με τις ψηφοφορίες μας και θα ξεκινήσουμε με το σημείο 27 θα ψηφίσουμε την έκθεση πρωτοβουλίας της Καριμά Ντελή. Έχετε την κάρτα σας όλοι. Θέλετε να κάνουμε μια δοκιμή πρώτα. μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ακούω κάποιους ήχους από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Υπότιτλος 1. Τροπολογία 61 δηλαδή. Του κυρίου Θέρκας. Η συγγήτρια είναι κατά υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 1. Συμβαστική τροπολογία D. Υπέρ. Κατά. Κλείσεις παρακαλώ πολύ τα τηλέφωνα. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρτη ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 21 ψήφοι υπέρ, 10 κατά, 3 αποχές. Επομένως εγκρίνεται η συμβαστική τροπολογία D. Επομένως καταπίπτουν κάποιες τροπολογίες και περνάμε συμβαστική τροπολογία ε από 5 πολιτικές ομάδες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Στην παράγραφο 1 πάντα, 71 τροπολογία της κυρίας Ζαμπόρσκα υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Στην παράγραφο 1 πάντα, τροπολογία 73 της κυρίας Τσούμπερ υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Στην παράγραφο 1 συμβαστική τροπολογία α μη την οποία έχουν υποβάλει τέσσερι πολιτικέ ομάδε υπέρ κατά αποχέ, εγκρίνεται. Στην παράγραφο 1 πάντα, τροπολογία 75 τη κυρία Τσούμπερ υπέρ κατά απόχέ, απορρίπτεται. 76 τη ίδια ηγήτρια, υπέρ κατά απόχέ, απορρίπτεται. παράγραφο 2, συμβασική τροπολογία F από τρει πολιτικέ ομάδε υπέρ κατά αποχέ. εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία AQ από τρεις πολιτικές ομάδες υπέρ AQ. Ναι, θα μπορούσαμε να το γράψουμε διαφορετικά. Έχουμε δύο γράμματα πάντως. AQ, υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος, αλλά νομίζω ότι απορρίπτεται. Άρτη ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 22 υπέρ, 16 κατά. Καμία αποχή. Επομένως εγκρίνεται. Τροπολογία 86 στην παράγραφο 2 του κυρίου Θέρκας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 3 συμβαστική τροπολογία G από 5 συγγνώμη διακόπτη πρόεδρος δεν έχετε διερμηνία εγώ μιλάω στα γαλλικά λογικά έπρεπε να υπάρχει διερμηνία προς τα αγγλικά Ωραία, λειτουργεί πολύ ωραία. Παράγραφος 3. Συμβαστική τροπολογία G από 5 πολιτικές ομάδες υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στη συμβαστική τροπολογία H από δύο πολιτικές ομάδες με μια προφορική τροπολογία από την εισηγήτρια. Υπάρχει κάποια ένσταση για την προφορική τροπολογία. Επομένως ψηφίζουμε τη συμβασική τροπολογία έτσι με την προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Στην παράγραφο 3 πάντα, τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Λοιπόν, τροπολογία 2 της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης υπέρ. Η συγκίτρια είναι κατά. Οι υπόλοιπε πολιτικέ ομάδε δεν γνωρίζω. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Στην παράγραφο 3, η 98 του κ. Νταρντέν υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 4, 3... Τροπολογίε για διαγραφή 102 τη κύρια Μακιντάιρ, 103 τη κυρία Τσίμερ και 104 του κυρίου Ομπερμάιερ. Θέλουν να διαγράψουν την παράγραφο 4 και οι 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Ψηφίζουμε τη συμβαστική ΑΗ από τρεις πολιτικές ομάδες υπέρ. Υπέρ της συμβαστικής τροπολογίας ΑΗ. Υπέρ παρακαλώ. Λοιπόν, ποιος είναι υπέρ της Συμβασικής τροπολογίας I, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 109 της κυρίας Τσούμπερ, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 110 της κυρίας Κλιβέτη, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 112 του κυρίου Σέρκας, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την 112 ζητάτε. Θα κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση λοιπόν. Νομίζω ότι μια πολιτική ομάδα δεν τα πηγαίνει πολύ καλά με αυτόν τον κατάλογο ψηφοφορία. Άρθρη ψηφοφορία για την 112. Ψηφίσατε όλοι πέρα. 19 υπέρ, 18 κατά, μία αποχή. Επομένω, η τροπολογία 112 εγκρίνεται. Παράγραφος 4 πάντα, συμβαστική τροπολογία J, από τέσσερις πολιτικές ομάδες υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. Παραγραφός 4, 116 από την εισηγήτρια, τον κύριο Μπένιον και τον κύριο Σέρκας υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 5, δύο τροπολογίες διαγραφής 117 και 118 από τους συναδέλφους Εσάγια και Ομπερμάιερ υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. Συμβαστική τροπολογία κάπα, την οποία έχουν υποβάλει Έξι πολιτικές ομάδες υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Γράφος 5. Τροπολογία 126. Τη συναδέλφου Γκαμπριέλε Τζίμερ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 128 της γήτρες και του φιλμπενιών υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 5, τροπολογία 131 της κυρία Τσίμερ υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Για τον υπότιτλο 1α, τροπολογία 133 του κύριου Νταρντέν υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Θα κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση για την 133. Άρτη ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 19 υπέρ, 20 κατά, καμία αποχή. Έχετε δίκιο λοιπόν, απορρίπτεται. Παραγράφος 5, τροπολογία 134 του κυρίου Νταρντέν με μία ενέτοιμα για χωριστή ψηφοφορία. Ψηφίζουμε το σύνολο του κειμένου χωρίς την φράση από το «Ergis Member States» έως «Partnership Contracts». Υπέρ τις 134 χωρίς το τμήμα το οποίο διάβασα. Κατά, αποχές, εγκρίνεται αυτό το πρώτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ της προσθήκης της φράσης αυτής. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται και αυτό. Παράγραφος 5 πάντα, τροπολογία 13 από την Επιτροπή Γυναικών υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 6. Συμβαστική τροπολογία L από 6 πολιτικές ομάδες υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 6. Τροπολογία ΑΚ από 3 πολιτικές ομάδες υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. Παράγραφος 7, 134, τροπολογία. 144, με συγχωρείτε, διορθώνει η Πρόεδρος. παράγραφος 7, τροπολογία 144 της κυρίας Τσουμπέρ, υπέρ. Κατά. Οι φιλελεύθεροι δεν ξέρω πώς ψηφίζουν, λοιπόν, 144 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 145 της, της κυρίας Μακιντάρη υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 8. Συμβαστική τροπολογία μη από 5 πολιτικές ομάδες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 8, 159 του κ. Ντερντέν υπέρ. 159 υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Παράγραφος 9, συμβαστική τροπολογία νη. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 9, 166 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 9 167 τροπολογία της κυρίας Αντζελίλη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 10 τροπολογία 168 για διαγραφή υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία ομικρών που έχει υποβληθεί από πέντε πολιτικές ομάδες υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 10. Συμβαστική τροπολογία π που έχουν υποβάλει πέντε πολιτικές ομάδες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 11. Συμβαστική Q υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 11. 181 της Εβελιν Ρέγνερ και του Βάντελ Χόλσερ υπέρ υπέρ λοιπόν κατά αποχές απορρίπτεται παράγραφος 11 συμβαστική R υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Παράγραφος 11, τροπολογία 184 του κυρίου Κοτσολίνο, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 12, τροπολογία διαγραφής 185 του Σόγκορ, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική S από τέσσερις πολιτικές ομάδες με, με ένα αίτημα προφορικής τροπολογίας. Υπάρχει κάποια ένσταση, όχι. Επομένως ψηφίζουμε την Συμβαστική τροπολογία S όπως τροποποιήθηκε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 12, τροπολογία 189 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 190 της συγγήτριας και του φιλμπενιών υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 12, τροπολογία 192 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 13, 193, τροπολογία διαγραφής του κυρίου Σόγκορ υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία ΤΑΦ από τέσσερις πολιτικές ομάδες υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 13, τροπολογία 197 της κυρίας Αντζελίλη υπέρ, κατά, αποχές Κοιτάξτε, ας κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση, άρτη ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρας. Κοιτάξτε, δεν αλλάζει τίποτα. 21 υπέρ, 6 κατά, 13 αποχές. Εγκρίνεται λοιπόν. Τροπολογία 198 της κυρίας Καστέξ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παραγράφος 14 συμβαστική γιού από δύο πολιτικές ομάδες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 15. Τροπολογία 213 για διαγραφή. Τροπολογία που έχει υποβάλει ο κύριος Σομπερμάιερ υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Μπορούμε να ψηφίσουμε τη συμβαστική Β από τρεις πολιτικές ομάδες υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 15, τροπολογία 218 του κ. Σόγκορ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 15, Τροπολογία 221 της ηγήτριας και του κυρίου Μπένιον με μία προφορική τροπολογία από την εισηγήτρια. Αν δεν υπάρχει ένσταση μπορούμε να ψηφίσουμε την τροπολογία υπέρ της 221. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 15 πάντα. Τροπολογία 223 του κύριου Πουπάκη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παραγράφος, ε, μάλλον τροπολογία 11 υπέρ, κατά αποχές, ας επαληθεύσουμε. Εάν ψηφίσατε όλοι, πέρας παρακαλώ. 21 υπέρ, 19 κατά. Απορρίφθεται. Α, δηλαδή εγκρίνεται, λέει η Πρόεδρος. Παράγραφος 16, συμβιβασμός W, τεσσάρων πολιτικών ομάδων, με προφορική τροπολογία, δεν διαφωνεί κανείς. Ψήφι υπέρ, λοιπόν, της W κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 16 τώρα έχουμε τη 267 υπέρ. Τι νονονο. Α, λάθος. Υπάρχει και άλλη συμβαστική προηγουμένως. ΑΠ. Συμβιβαστική στη σελίδα 22. Είναι μια συμβαστική τροπολογία που αφορά πάντα την παράγραφο 16 και έχει καταδεθεί από τρεις πολιτικές ομάδες. Ψήφι Κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα θα πάμε στην 267 της κυρίας Κλειβέτη μετά την παράγραφο 16. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 16 πάντα η 269 της εισηγήτρια και του κυρίου Σέρκας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 9 της Επιτροπής Γυναικών Α, όχι, θα ψηφίσουμε το συμβασμό Α, Ναι. Βάλαμε μπρος τη μηχανή του χρόνου. Έξι πολιτικών ομάδων. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα, στην 9 τη επίτροπή Γυναικών υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2.71 της εισηγήτρια και του Φιλμπένιον υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2,73 εισηγήτριας υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2,74 της ιδίας υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2,75 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3 τη Επιτροπής Γυναικών υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 17. Συμβασμός X υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, μετά την παράγραφο 17 η 9 της Ρέγγι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 282 μπένιον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 283 της αντιπρόεδρου μας κυρία Σούμπερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.85 Μπένιον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.86 Τσάμπα Σόγκορ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.87 Άννα Ζαμπόρσκα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.88 της εισηγήτρες και του Μπένιον με προφορική τροπολογία διαφωνεί κανείς όχι ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μετά την παράγραφο 17 συμβασμός Α.Ε.Λ. 5 πολιτικών ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 10 Επιτροπή Γυναικών υπέρ κατά, όχι παράγραφος, τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.91 εισηγήτρια υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 5 Επιτροπής Γυναικών υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Στην παράγραφο 18-293 του Τσάμπα Σόγκορ για διαγραφή υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ψηφίζουμε τη 294 της ηγήτρας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 19 συμβασμός Υ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 20 συμβασμός ΑΑ τριών ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 20 συμβασμός ΑΒ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 20 τροπολογία 3.14 μπαίνουν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3.15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3.16 του Μπένιον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μετά την παράγραφο 20 πάντα 3.17 της ηγητρίας με προφορική τροπολογία της Ιδίας διαφωνεί κανείς Ψηφίζουμε. Ψήφι υπέρ της 317 όπως τροποποιήθηκε. Κατά αποχές εγκρίνεται. 318 εισηγήτρια και μπένιον υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 319 των ιδίων υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 21. Δύο τροπολογίες προς απαλληψη 3.23.21, 323-21. Μάκιντάιρ και Σόγκορ. Ψηφίζουμε. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 322 Ψάρι Εσαΐα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3.23 της εισηγήτριας συμβατή υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τώρα αιτιολογική αναφορά 1 υπέρ της τροπολογίας 1 κατά απόχέ. εγκρίνεται της εισηγήτριας τροπολογία 2 3 και 4 Σέρκας, Καστέξ και Ρέγνερ και Βάιντεν Χόλτσερ ταυτίζονται και τις ψηφίζουμε ομού 2-3-4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται <clears throat> αιτιολογική αναφορά 2 η, τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συγγνώμη. μετά έχουμε την 6 Καστέξ Σέρκας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 δεν το ψηφίζουμε. Μετά την αιτιολογική αναφορά 24, η 8 της ηγήτρε υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Μετά έχουμε το συμβιβασμό α τριών πολιτικών ομάδων υπέρ κατά απόχέ. εγκρίνεται. Μετά την 37 έχουμε την 11 τροπολογία Σέρκας και Καστέξ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 12 της κυρίας Κοστέλο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την αιτιολογική αναφορά 43, η τροπολογία 15 του κυρίου Κοτσολίνο και του κυρίου Καρόνα. Υπέρ. Contre abstention. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 16 της κυρίας Τσίμερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 17 κοτσολίνο είπε. κατά αποχές εγκρίνεται η αιτιολογική σκέψη α η τροπολογία 18 Φρανς Ομπαμάια α είναι για διαγραφή είπε. κατά αποχές απορρίπτεται άρα ψηφίζουμε το συμβασμό α που έχουν καταθέσει πέντε ομάδες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μετά την αιτιολογική σκέψη α, έχουμε ένα συμβασμό αε, πέντε πολιτικών ομάδων υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά την αιτιολογική σκέψη α πάντα, νέος συμβασμός ΑΣΕ Των ιδίων πέντε πολιτικών ομάδων υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη Β, συμβιβασμό Β, έξι πολιτικών ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Στη συνέχεια, πάντα στην αιτιολογική σκέψη Β, παράγραφο Σ τη Επιτροπή Γυναικών υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάντα στην ίδια αιτιολογική σκέψη Β, συμβιβαστική τροπολογία ΑΕΦ τριών ομάδων υπέρ κατά αποχές υπέρ παρακαλώ ΑΕΦ συμβιβαστική τροπολογία κατά Αποχές εγκρίνεται. Πάντα στην αιτιολογική σκέψη Β, Α, Ή. Πέντε πολιτικές ομάδες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ο συμβιβασμός. Πάντα στην ίδια αιτιολογική σκέψη συμβασμός AG των ιδίων πέντε ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάντα στην ίδια σκέψη, παράγραφος ΔΕΛΤΑ Επιτροπή Γυναικών υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάντα στην αιτιολογική σκέψη Β, συμβασμό ΑΔ, πέντε πολιτικών ομάδων. Υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Πάντα στην αιτιολογική σκέψη Β, η τροπολογία 37 του Αλεχάνδρου Σέρκα υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη Γ, συμβασμό σε, τεσσάρων ομάδων υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Μετά του ΣΕ, η τροπολογία 46 συγκήτριας Μπένιον και Σέρκας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 47, Γκαμπριέλ Τσίμερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 48, Νταρντέν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 49, Κόστελο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την αιτιολογική σκέψη σε, η συμβαστική, αχ, εδώ, α, ή, τεσσάρων πολιτικών ομάδων υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη C, AG, ε, συμβιβασμός υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά την αιτιολογική σκέψη σε παράγραφος είτε επιτροπή Γυναικών, η συγκίτρια είναι αντίθετη υπέρ κατά Ξανά. Πάμε από την αρχή. Επιτροπή Γυναικών, έτσι. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε έλεγχο. Ας το ελέγξουμε λοιπόν. Άρχεται η παλήθευση. Ψηφίζουμε την παράγραφο H της Επιτροπής Γυναικών με την εισηγήτρια κατά. Εάν ψηφίσατε όλοι πέρας. 28 υπέρ, 22 κατά. Δεν εγκρίνεται λέει η Πρόεδρος τώρα. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται η ΚΕΙΕΝ. Η 55 σήμερα. Έλεγχο θέλετε. Ωραία, εντάξει, εντάξει. Είναι μικρή η διαφορά, το ελέγξουμε. Tout le monde a pu voter, Ψήφισατε όλοι. 24 υπέρ 18 κατά, χωρίς αποχές, εγκρίνεται. Είχατε δίκιο που ζητούσατε θέση. Ή 55 τσίμερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται σαφώς. Και ερχόμαστε στην τροπολογία 57 της κυρία Τσίμερ και πάλι ψήφι κατά αποχές αποχές εγκρίνεται και τελειώσαμε περίπου έχουμε την τροπολογία 60 του κυρίου Νταρδέν. Φρεντερίκ υπέρ. τα αποχές εγκρίνεται σαφώς. Ψηφίζουμε λοιπόν το σύνολο της έκθεσης πρωτοβουλίας ηλεκτρονικά όπω τοποποιήθηκε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. «26 υπέρ, 3 κατά, 16 αποχές». Συγχαρητήρια κυρία Συγκήτρια. Και τώρα Πάμε στο σημείο 23. Κάντε λίγη ησυχία σας παρακαλώ. Θα ψηφίσουμε τη γνωμοδότηση του συναδέλφου Ζόρζ Μπαχ της Επιτροπής Αερομεταφορών αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων στην εξωτερική πολιτική αερομεταφορών. Μετά την παράγραφο 1 έχουμε την τροπολογία 3 του εισηγητή υπέρ Κατά αποχές εγκρίνεται. 4 του ιδίου υπέρ. Κατά αποχές το ίδιο. 5 το αυτό υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 6 του ιδίου υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 7 του ιδίου υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 8 κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 1, πάντα συμβαστική α, δύο πολιτικών ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 2, παρά 11 τροπολογία του εισηγητή. Ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 2, 14 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και πάλι συμβαστική ε, μπέ, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ναι. Παράγραφος 3, η τροπολογία 15 υπέρ της κυρία Στάιρου κατά αποχές εγκρίνεται. Η 16 της ιδίας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 4-17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 18 της ιδίας υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές. είπα. κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 4, 19 με προφορική τροπολογία που βλέπετε εδώ, σοσιαλιστές και δημοκράτες, δεν διαφωνεί κανείς. Ψηφίζουμε λοιπόν όπως τροποποιήθηκε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 4, τροπολογία 20 της ιδίας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 5, συμβασμό σε πολιτικών ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την 5, 23 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 24 της ηγήτρες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 25 της ιδίας κατά του ιδίου, συγγνώμη, 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 27 του κυρίου Μπαχ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 28 Μπαχ 20, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την αιτιολογική σκέψη α, μια ανθρωπολογία 1, της κυρία Στάιρουκ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Οι δύο, της ιδέας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το σύνολο της γνωμοδότησης θα ψηφίσουμε τώρα η ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Έληξε. 35 υπέρ, 5 κατά μία αποχή. Συγχαρητήρια. Και είναι 35. Στο 24 ψηφίζουμε ψηφίζουμε την έκθεση Μορέν Σαρτιέ για τη συμφωνία με το Συμβούλιο σε πρώτη ανάγνωση για την οδηγία με τους εργαζόμενους που εκτίθενται σε σωματικούς κινδύνους και ιδιαίτερα ηλεκτρομαγνητικά πηδία. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά όπως συμφωνήθηκε με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 26 Μαρτίου και συμφώνησε από αυτού 10 Απριλίου και το Κορεπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι, έληξε 38 ψήφοι υπέρ, 2 κατά, καμία αποχή. Συγχαίρουμε την εισηγήτρια. και τη διαπραγματευτική ομάδα. Και, και τώρα το 25. Έκθεση πάλι της κυρίας Μωρέν Σαρτιέ για την τροποποίηση της πρότασης της Κομισιόν προς τον κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ώστε να συμπεριληφθεί και η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. 3-1-α ή συμβιβαστική Β, από πέντε ομάδες, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 5-1-β, τροπολογία 5, των κυριών Σρόντερ και Μωρέν Σαρτιέ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 15 Ι υποπαράγραφος 1 συμβιβαστική γάμα από τέσσερις ομάδες. Δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε. Χρειάζεται, χρειάζεται να ψηφίσουμε. Τα διάβασα ανάποδα λέει η Πρόεδρος. Λοιπόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 15 υπό υποπαράγραφος 2 νέο σημείο από τέσσερις ομάδες συμβαστική α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μετά το 15 γιώτα, τροπολογία 12 του Πολ Μάρφη Ινιές Χριστίνα Σούμπερ και Πατρίκ Λεϊαρίκ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 15 Ρωμαϊκό μικρό 3 υποπαράγραφος 2α τροπολογία 13 Ελισάβετ Σρόντερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 άρθρο 15 Ρωμαϊκό μικρό 4 παράγραφος 1 συμβιβαστική 4 τεσσάρων ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15-5 τροπολογία 18 της ΓΚΟΕ για διαγραφή υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Στην προσθήκη 2 παράγραφος 2 1 τροπολογία 19 του Αλεχάνδρου Σέρκας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προσθήκη 2 παράγραφος 2 σημείο 1 α νέο τροπολογία 20 της κυρίας Μωρέν Σαρτιέ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 21 του Αλεχάνδρου Σέρκα, υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 22 τη εισηγήτριας υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Στη προσθήκη 2 παράγραφο 2 σημείο 3 τροπολογία 23 του Αλεχάνδρου Σέρκα υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 24 τη εισηγήτριας υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβιβαστική ε, τεσσάρων ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 27 της ΓΟΕ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 τροπολογία των ιδίων υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 29 έχει καταπέσει. Ψηφίζουμε τώρα μετά το σκεπτικό γάμα. Α, όχι, όχι, αυτό καταπέσει. Εγκρίναμε λοιπόν την τροποποίηση του κανονισμού και η τροποποίηση αυτή του κανονισμού θα μπει μέσα στην εντολή, στη διαπραγματευτική εντολή που αποτελείται από μια γυναικεία Dream Team. Τελείωσε και αυτό το σημείο και τώρα πάμε στην ψήφιση ενός κειμένου σχετικό με τα προηγούμενα, στο σημείο 26 δηλαδή της ημερήσιας διάταξης. Τροπολογίες στο σχέδιο κανονισμού, κοινού κανονισμού για τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία και άλλα. Και ο εισηγητής, γιατί ο συντάκτης μάλλον είναι ο συνάδελφός μας Αδάμ Κόσα. Είναι γνωμοδότηση προς την Περιφερειακή Επιτροπή. Άρθρο 18, δύο τροπολογίες για διαγραφή, 4 και 5 του Αλεχάνδρου Σέρκας και του εισηγητή. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Άρθρο 83, παράγραφος 1, τροπολογία 6 του Αλεχάνδρου Θέρκας και της Ελισάβετ Μορέν Σαρτιέ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. τροπολογία 7 χωρίς όμως τους αριθμούς υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται άρθρο 83 παράγραφος 2 τροπολογία 8 της ΓΚΟΕ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται άρθρο 84 παράγραφος 3 α τροπολογία 9 δεν μπορεί να ψηφιστεί, να παράδεκτη Ψηφίζουμε όμως την τροπολογία 10 του Αλεχάνδρου Θέρκας και της Ελισάβετ Μορέν Σαρτιέ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 84 παράγραφος 3 β. Νέα. Τροπολογία 11 του Αλεχάνδρου Σέρκας υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Προσθήκη 3 3. Παράγραφος 1. Συμβιβαστική α2 ομάδων. ΕΛΚ και σοσιαλιστές. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προσθήκη 5. Τροπολογία 15. Διαγραφής από την ΓΚΟΕ. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική β των δύο ιδίων αυτών ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική γ των δύο ιδίων ομάδων αυτών υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά το σκεπτικό 57, τροπολογία 1 του Αδάμ Κόζα και της Ελισάβετ Μωρέν Σαρτιέ. Α, όχι, προηγουμένως πρέπει να ψηφίσουμε την τροπολογία 20 του Αλεχάνδρου Σέρκας γιατί δεν εγκρίθηκε η 15. Η τροπολογία 20 λοιπόν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τώρα μετά το 57, εγώ σκεπτικό 57, τροπολογία 1 του ΑΔ. Τι θέλετε κύριε Πριότο να παρέμβετε. Ναι, Πρόεδρε, σε αυτήν την αιτιολογική σκέψη έχω μια προφορική τροπολογία να κάνω. Στο τέλος της δεύτερης παραγράφου, μια στιγμή περιμένετε, λέει ναι. Πρόεδρος, να το βρω. Κουλ, κουλ, κουλ. Βρήκατε, ναι. Λοιπόν, λέω, στο τέλος της δεύτερης παραγράφου να προσθέσουμε το εξή κείμενο. Η εγγύηση για την απασχόληση των νέων θα πρέπει να υποστηρίξει νέους χωρίς εργασία, ε, μόρφωση ή κατάρτιση ε, που ε, είναι στις επιλέξιμες περιφέρειες και μέσα σε ένα τετράμινο μετά τη λήξη της μαθητείας τους. Το ίδιο είχαμε γκρίνει στην έκθεση της κυρίας Μωρέν Σαρτιέ στο συμβιβασμό Α. Είναι ακριβώς το ίδιο κείμενο. Και το έχουμε βάλει και στο συμβιβασμό την περασμένη εβδομάδα στη συνεδρίαση των σκιωδών εισηγητών. Γιατί υπάρχει ένα ασφάλμα του κυρίου Κώσα, χρειάστηκε να φύγει από τη συνεδρίαση ε, των σκιωδών και τώρα ε, δεν είναι ο συμβασμός αυτός ε, ε, στη λίστα ψηφοφορία. Δεν μπορέσαμε να βρούμε τον κύριο Κώσα για να του συζητήσουμε μαζί του, αλλά πολιτικά έχουμε συμφωνήσει. Γιατί ο στόχος είναι να είναι παράλληλες εκθέσεις και ε, συνεκτικές και ε, συναφεί μεταξύ του Γι' αυτό και η προφορική τροπολογία. Ναι. Αλλά αυτό που λέτε είναι στην τροπολογία 2. Ενώ ψηφίζουμε την τροπολογία 1. Άρα, υπέρ τη 1, χωρί προφορική. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Για την τροπολογία 2 υπάρχει καμία αντίρρηση στην προφορική τροποποίηση που μόλι προτάθηκε. Όχι, λοιπόν, ψηφίζουμε την τροπολογία 2 με την προσθήκη υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 3 είναι συμβατή του Πολ Μόρφη και του Πατρίκ Λεγιαρίκ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελείωσε και αυτό το σημείο. Θα συμπληρωθεί και αυτό θα συμπεριληφθεί στη διαπραγματευτική εντολή που είναι και αυτή από Dream Team. Dream Team αλλά όχι γυναικεία. Τελείωσε, τελείωσε λέγω, τελείωσε. η ψηφοφορία. Σιωπή παρακαλώ. Τώρα το 13 όμως θα δώσω το λόγο στο συνάδελφό μας Θωμά Χέντελ για να μας παρουσιάσει το σχέδιο έκθεσης πρωτοβουλίας του για τις διαπραγματεύσεις, για τις διαμεθοριακές διαπραγματεύσεις και τον κοινωνικό διάλογο είναι το σημείο 13 της ημερήσιας διάταξης. Κύριε εισηγητά, θα πάρετε το λόγο μόλις λήξει ο θόρυβος. So, vielen Dank, Frau ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς, θα πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Οι συνάδελφοί μου του Συνδικάτου Βέρντι στη Γερμανία ε, με εμπόδισαν να παρουσιάσω γέρο σήμερα την έκθεσή μου ε, σκόνταψα ε, στην απεργία της Λουφτχάνσα και έφτασα μόλις σήμερα στις Βρυξέλλες. Είναι πραγματικά ευτράπελο αυτό στη συγκεκριμένη έκθεση. Ε, λοιπόν, την έκθεση αυτή την έχουμε συζητήσει και σε hearing, σε μια δημόσια κρόαση. Είδαμε τις διάφορες επεκτάσεις και επιπτώσεις που υπερβαίνουν κατά πολύ το πλαίσιο της έκθεσης της ίδιας. Τώρα, για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις, Μήπως έξω τα πηγαδάκια, συνάδελφοι, και οι ε, Θα ήθελα λοιπόν να προεξοφλήσω κάτι. Περί δεν πρόκειται. Καλά, έτσι κι αλλιώς δεν είναι κανείς εδώ και αυτοί που είναι εδώ μιλάνε. Λοιπόν, ήθελα να προεξοφλήσω ε, ευθύ εξ αρχή, Γιατί δεν έχω βάλει διάφορα πράγματα που μου ζητάνε διάφοροι σκιώδεις συγητές διαφόρων πολιτικών ομάδων. Τι θέλει αυτή η έκθεση. Δεν ασχολείται με το θέμα του μισθού τι συλλογικέ διαπραγματεύσει για τι συμβάσει, ούτε καν για ένα ευρωπαϊκό συντονισμό για το μισθό. Καμία σχέση όλα αυτά. Ε, τι θέλουμε εμεί. Μάλλον κάτι άλλο που δεν θέλουμε είναι οι συλλογικές συμβάσεις. Αυτό, ε, υπάρχει αυτονομία στα κράτη-μέλη. Ε, ε, είναι και συνταγματικού χαρακτήρα και αλλήμον εάν ανοίγαμε αυτούς τους ασκούς του αιώλου σε μια τέτοια έκθεση και ούτε κάνουμε μισθό συντονισμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίσης δεν φύγουμε την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων που ε, είναι θεμελιώδες το δικαίωμα για τις συλλογικέ διαπραγματεύσεις στην Ευρώπη. Όλα αυτά λοιπόν δεν είναι αντικείμενο της έκθεσης. Την έκθεση αυτή την ανέλαβα αργά. Δεν την ε, προκαλέσαμε εμείς αυτή την έκθεση. Έχει μακρά προϊστορία ετών, για να μην πω δέκα ετιών, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μελέτες επιμελετών, τόμοι ολόκληρη, χοντρά βιβλία. Τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δραστηριοποιήθηκε και πάλι και προσπαθεί ε, κάπως να προχωρήσει αυτό το θέμα. Και χρειάστηκε να γνωμοδοτήσουμε και εμείς. Πάρα πολύ γρήγορα να σας εξηγήσω λοιπόν το έγγραφο. Πρώτον, αυξάνονται όλο και περισσότερο οι διεθνείς συμφωνίες, οι διασυνοριακές στην Ευρώπη. Και επιταχύνονται κιόλας ενώ τις διμερείς, έτσι, όχι τις διεθνείς, τις συμφωνίες μεταξύ των διαφόρων κρατών, διακρατικές. Δεύτερον, προτείνω στην έκθεση αυτή μια εθελοντική ή προαιρετική μορφή νομικού πλαισίου που μέχρι σήμερα δεν υπάρχει. Μου είπανε ότι μάλλον πάνε καλά τώρα, τι θέλεις και τα ανακατεύεις. Άκουσα όμως πολλές περιπτώσεις τέτοιων διεθνών συμφωνιών σε επίπεδο επιχειρήσεων, όπου όμως αυτές δεν τηρήθηκαν από το ένα συμβαλόμενο μέρος. Ε, γι' αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να ε, δημιουργήσουμε τέτοιο νομικό νομοθετικό πλαίσιο, εθελοντικό, για να υπάρχει κάποια στοιχειώδης ασφάλεια όταν ε, συνάπτουν τέτοιες συμφωνίες. Τρίτον, επειδή είναι και διαφορετικές οι δομές εκπροσώπησης συμφερόντων, κατά την άποψή μου θα πρέπει να δώσουμε στα ευρωπαϊκά συνδικάτα μια ισχυρή εντολή. Και τα ευρωπαϊκά επιχειρησιακά συμβούλια δεν είναι υποκατάστατα ε, των διαπραγματεύσεων. Δεν πάνε έτσι οι διάφορες δομές συγκρότησης συμφερόντων στην Ευρώπη. Θα ήθελα όμως να πω ότι τα Ευρωπαϊκά Επιχειρησιακά Συμβούλια θα πρέπει να συμμετέχουν ε, σε αυτή την ομάδα. Και βάσει λοιπόν ε, των περιπλοκών θα πρέπει να υπάρχουν και μηχανισμοί εξοδικαστικής επίλυσης διαφορών. Όταν κάποιος έχει συνάψει μία σύμβαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ε, διακανονισμού εξοδικαστικής μορφής όταν κάποιος δεν τηρεί τις αρχές και όχι ε, σύμφωνα με τη συνθήκη της Ρώμης 1 γιατί αυτές είναι ιδιωτικά συμφωνητικά και τέτοιες ε, συμφωνίες δεν έχουν να κάνουν με συλλογικά δικαιώματα. Και επίσης θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει και μια ευρωπαϊκή υπηρεσία επίλυσης διαφορών σε επίπεδο, ας πούμε, εργατοδικείο, γιατί υπάρχουν ε, κάποια θέματα που αν πρέπει να φτάνουν στα δικαστήρια δεν είναι αρμοδιότητα του σημερινού Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ένα τέτοιο λοιπόν πλαίσιο ε, θα πρέπει να ε, αφορά συλλογικά μέτρα με διασυνορική εφαρμογή. Ε, με βάση τη σημερινή νομολογία και τις ανασφάλειες που υπάρχουν, δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι αυτά θα μένουν εκτός ενός ενιαίου πλαισίου επίση καλωσορίζουμε τι δραστηριότητε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των διαφόρων κοινωνικών εταίρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με ενημέρωση και συνεχείς διαβουλεύσεις. Όλα αυτά θα πρέπει να μετεξελιχθούν, να αναπτυχθούν και τελικά ε, να βοηθήσουν να προχωρήσει έτσι περαιτέρω ο ευρωπαϊκός κοινωνικός διάλογος. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και με χαρά περιμένω τις συζητήσεις που πραγματικά θα είναι ενδιαφέρουσες πιστεύω. Monsieur Oui Σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την έκθεσή του αυτή. Εν γέννη συμφωνώ με την προσέγγισή του το ότι θα πρέπει να είναι αυτόνομη η κοινωνική εταίρη. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε και μία ρήτρα που να αποτρέπει αρνητικές επιπτώσεις στις εθνικές συμφωνίες. Και κατά αυτόν τον τρόπο θα βελτιωθεί και ο κοινωνικός διάλογος. Αυτό δεν υπονομεύει σε καμία περίπτωση βέβαια τις εθνικές συλλογικές συμβάσεις και νομίζω θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και κάποιες από τις συμβάσεις της Διεθνής οργάνωση Εργασίας, να τις αναφέρουμε δηλαδή στην αιτιολογική σκέψη και να χρησιμοποιήσουμε επίσης και τη σύμβαση του ILO, τη Διεθνής, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, ως ελάχιστη βάση για τις εργασιακές αυτές συμβάσεις. Δεν ξέρω όμως ε, πώς θα καταφέρουμε να συνδυάσουμε με όλα αυτά τα οποία λέγονται εδώ πέρα, τα δικαστήρια τα αρμόδια για την επίλυση των δικαστικών εργασιακών διαφορών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως μας λέει ο εισηγητής, επί του παρόντος, δεν μπορούμε ακόμα να εγκρίνουμε μέτρα διασυνοριακής επίλυση εργασιακών διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι μπορούν ακόμα και οι νομοθεσίες να επηρεάσουν πάρα πολύ τον τρόπο με τον οποίο εκδικάζονται κάποιες υποθέσεις, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αν δεν έχουμε ξεκάθαρους κανόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε μπορούμε να έχουμε και πολλές διαφορετικές δικαστικές αποφάσεις για την ίδια δικαστική διένεξη, για την ίδια δικαστική διαφορά, πράγμα το οποίο πρέπει να αποφύγουμε. Πρέπει δηλαδή να μπορούμε να σε θέση να προβλέψουμε λίγο την έκβαση μιας διαφοράς και βέβαια αν καταλήξουμε σε κοινέ συμφωνίες ότι θα πρέπει να μπορούμε να έχουμε και ένα κοινό σύστημα επίλυσης των διαφορών που μπορούν να προκύψουν σε σχέση με μια τέτοια συμφωνία ή σύμβαση. Θα ήθελα λοιπόν να συζητήσουμε περισσότερο το ζήτημα αυτό με περισσότερε λεπτομέρειε. Για μένα είναι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή, στα πλαίσια αυτή τη έκθεση πρωτοβουλία, να εντοπίσω μια λύση. Είναι πολύ σημαντικό να υποστηρίξουμε του κοινωνικού εταίρου, να εξελιχθεί περισσότερο ο κοινωνικό διάλογο και υπάρχουν και ορισμένοι τομεί που θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν καλύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπω είπε πάντω ο εισηγητή, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να διασφαλίσουμε την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων. Αυτοί θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι για τα ζητήματα που εξετάζουμε. Αυτοί θα πρέπει να αναπτύσσουν τα διάφορα εργασιακά μοντέλα. Πρέπει εμεί όμως με κάποιο τρόπο, μέσω συγκεκριμένων κανόνων, να τους υποστηρίξουμε και να δώσουμε μεγαλύτερη διαφάνεια σε κάποιου τομεί, όπως για παράδειγμα επαγγελματική κατάρτιση. Προσβλέπω πάντως στη συνέχεια της συζήτησης και ελπίζω θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα που πραγματικά θα βοηθήσει τις συνδικαλιστικές οργανώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ελπίζω ότι θα καταφέρουμε τελικά να τις βοηθήσουμε να αυξήσουν την επίδρασή τους. Η κυρία Σρέντερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ενδιαφέρουσες οι προτάσεις αλλά επειδή δεν είχαμε και χρόνο, είναι επιγραμματικά τα περισσότερα. Εγώ σαν τον συνάδελφο Λούτβιξον έχω καμιά χιλιάδα ερωτήματα που ανακύπτουν. Κάπου που θα πρέπει να έχουμε ένα μπούσουλα, ένα στόχο. Έχουμε μια εφιστάμενη κατάσταση συνθήκων, δεν μπορούμε να ζητάμε πράγματα, τον ουρανό μετάστρα πέρα από τη συνθήκη έχουμε ένα πλαίσιο που μας περιορίζει. Και επιθυμούμε τροποποίηση με των συνθήκων, να το πω δεύτερον. Λαμβάνεται πολύ λίγο υπόψη ότι υπάρχουν πολύ διαφορετικές εθνικές παραδόσεις ως προς το ρόλο των κοινωνικών εταίρων και αυτό παίζει μεγάλο ρόλο. Αλλιώ δεν θα βρούμε πλειοψηφία όσο καλές και αν είναι οι διατυπώσεις διακυβεύονται σε ορισμένα κράτη πράγματα που θεωρούνται αυτονόητα και συνταγματικά, ιδιαίτερα για την επίλυση των διαφορών, έχω επιφυλάξεις και αμφιβολίες. Μετά, σε ποιο πλαίσιο θα γίνονται αυτές οι συμβάσεις, το ξέρω ότι υπάρχουν, αλλά σε ποιο βαθμό θα πρέπει να διευρυνθούν, είναι για μένα ένα ερώτημα αυτό, και επίσης ποιους εργαζομένους αφορά αυτό άνδρες και γυναίκες, τις κλασικές μορφές. Μα δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Έχουμε δυσκολία διεθνώς. Έχουμε συνθήκες απασχόλησης και σχέσεις εργασιακές που ξεφεύγουν από κάθε γνωστό πλαίσιο. Αυτό δεν το λέει η έκθεση. Και νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να προτείνει το Κοινοβούλιο. Το πιο σημαντικό για μένα δεν αναφέρεται καθόλου. Είναι ή διασυνοριακές κλασικές διαπραγματεύσεις που, βρίσκ, που είναι και παραμεθόριες και έχουν μια πολύ ε, ιδιαίτερη περιφερειακή διάσταση. Έχουν και ένα ευρωπαϊκό στοιχείο και ευρωπαϊκή λειτουργία πέρα από τα ευρωπαϊκά επιχειρησιακά συμβούλια. Στις παραμεθόριες περιοχές είναι πάρα πολύ σημαντικό οι κοινωνικοί εταίροι να καταλήγουν σε διαπραγμάτευση και επίσης κάτι άλλο που λείπει από την έκθεση είναι τι γίνεται με τις διαπραγματεύσεις ε, για τους μισθούς. Τις ευρωπαϊκές υπάρχουν πέρα από τις εθνικές αναπτύσσονται στρατηγικές, γίνονται συνεργασίες, αλλά θα πρέπει να το συζητήσουμε οι σκιώδες συζητητές και να εμβαθύνουμε περισσότερο σε αυτά τα ζητήματα και σε αυτή τη στρατηγική. Γιατί αυτό είναι ακριβώς αυτό που μας ενδιαφέρει. Στα πλαίσια μιας έκθεσης πρωτοβουλίας μπορούμε να κάνουμε προτάσεις, το είδαμε στην εγγύηση για την απασχόληση των νέων. Θα πρέπει όμως να συμφωνήσουμε για κάτι εφικτό και όχι να έχουμε υπερβολικές απαιτήσει και να συγκρουστούμε με συντάγματα. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να δούμε τι γίνεται πραγματικά στα σύνορα, στις περιφέρειες που χρειάζεται ρύθμιση, γιατί υπάρχουν ε, εργαζόμενοι που ζουν σε μια χώρα και δουλεύουν στη διπλανή. Εκεί είναι το μεγαλύτερο κοινωνικό ντάμπινγκ. Αυτό επίσης έχει να κάνει και με τους κλάδους ε, μέρους. Πώς να το πω. Υπάρχουν και νοικιαζόμενοι, αποσπασμένοι εργαζόμενοι. Με αυτούς τι γίνεται. Υπάρχουν ειδικές συμβάσεις, ιδιαίτερες πλέον στην Ευρώπη, και είναι δύσκολο να διαχειριστεί κανείς αυτά τα θέματα γιατί δεν ξέρουμε τελικά τι ρόλο παίζουν εκεί ε, όλα αυτά τα φαινόμενα ή είναι οι κλασικές μορφές και σχέσεις εργασίας, εργαζόμενοι εργοδότες. Θα ήθελα πάρα πολύ να το συζητήσουμε στην ομίγυρη των σχεδόν εισηγητών εντατικά για να καταφέρουμε ένα σαφές πλαίσιο και να μην ζητάμε πάρα πολλά πράγματα. Γιατί κρίμα, θα πάει στο βρόντο αυτή η πρωτοβουλία και δεν θα υπάρχει μεγαλύτερη κοινωνική εξασφάλιση των εργαζομένων, πράγμα που θέλουμε εμείς κυρία Κορνέλησεν. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι έρχεται την κατάλληλη στιγμή αυτή η έκθεση. Και είναι σημαντικό να την αντιμετωπίσουμε σφαιρικά. Έχουμε το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, την οικονομική διακυβέρνηση που έχει προστεθεί τώρα και που αρχίζει και ασχολείται και λίγο με την κοινωνική πολιτική και την απασχόληση και όπου βλέπουμε ότι υπάρχουν όλο και μεγαλύτερες μακροοικονομικές ανισότητες ως προς τον τομέα αυτό, δηλαδή της απασχόλησης. Ενώ βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν διεθνοποιήσει πλέον τη δραστηριότητά τους, έχουν γίνει πιο διεθνείς και βλέπουμε ότι οι εργαζόμενοι, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, τα συμφέροντά τους υπολείπονται πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ εθνικά ακόμα. Επομένως, έχουν χάσει πάρα πολύ την εξουσία τους πλέον, τη δύναμή τους, περιορίζονται μόνο σε εθνικό επίπεδο. Και αυτό που βλέπουμε είναι ότι είμαστε όλο και πιο διασυνδεδεμένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει λοιπόν να βρούμε τρόπους για να ανακτήσουμε κάπως τη δύναμη του κοινωνικού διαλόγου σε ευρωπαϊκό επίπεδο και για να δώσουμε μεγαλύτερη ισχύ στι συλλογικέ διαπραγματεύσει, ιδίω σε αυτή τη χρονική στιγμή που το Συμβούλιο πρόκειται να εξετάσει την κοινωνική διάσταση τη Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι αυτή η κατάλληλη στιγμή για να σκεφτούμε κι εμεί πολλού τρόπου για να εκδημοκρατήσουμε το ευρωπαϊκό εξάμεινο και να δώσουμε έναν πιο διεθνικό ρόλο στον κοινωνικό διάλογο. Η Νάντια Χίρισε έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την έκθεσή του. Και μαζί με τον συνάδελφο Κρόιτσμαν είμαστε σκιώδεις εισηγητές για την έκθεση αυτή. Οι φιλελεύθεροι έχουν βάλει δύο σκιώδεις εισηγητές. Χαιρόμαστε για τη συζήτηση. Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και ο διασυνοριακός διάλογος θα προσλαμβάνω όλο και περισσότερο σημασία στο μέλλον, ακόμα και αν είναι περιορισμένοι σε αριθμό σήμερα αυτοί οι εργαζόμενοι, αλλά είναι ακόμα ένα ορόσημο και ένα λιθαράκι για να ολοκληρωθεί η ενιαία αγορά. Και για μας τους φιλελευθέρους είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κοιτάξτε, με αυτή, την Μάλλον με αυτή την πρωτοβουλία δεν θα πρέπει να αυξήσουμε τη γραφειοκρατία ακόμα περισσότερο, να το προσέξουμε και να δούμε πού ταιριάζει να χρησιμοποιείται. Αυτός ο προαιρετικός χαρακτήρας του πλαισίου είναι πολύ σημαντικό να παραμείνει προαιρετικός. Έχουμε κάποια ερωτηματικά εμείς για την εξοδικαστική επίλυση των διαφορών. Τι είναι αυτό? Μήπως υπερβάλλουμε για αυτή την τριμερή μορφή που προτείνεται πρέπει οπωσδήποτε να γίνει. Για όλες αυτές τις ρήτρε που προτείνεται να συμπεριληφθούν στις ε, διαπραγματεύσεις, μήπως είναι καλύτερο να επενδύουμε στην εμπιστοσύνη ε, στη σχέση των εργαζομένων με τους εργοδότες. Πάντως, περιμένουμε με μεγάλη χαρά και ανυπομονησία τη συζήτηση. Θα είναι ενδιαφέρουσα η έκθεση. Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ. Να πω και εγώ κάποια λόγια. Όντω η συζήτηση αυτή γίνεται την κατάλληλη στιγμή, μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για πολλού λόγου. Καταρχάς, νομίζω ότι θα πρέπει να ενημερώσουμε τα μέλη της Επιτροπής μας, για όσους δεν το γνωρίζουν, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να μην δώσει συνέχεια στην έκθεση νομοθετικής πρωτοβουλίας, την οποία συντάξαμε, όσον αφορά την υπευθυνότητα, έκθεση του κυρίου Σέρκας, μάλλον με συγχωρείτε, έκθεση του κυρίου Σέρκας όσον αφορά την αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων. Ξέρετε ότι η απόφαση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ελήφθη χωρίς να προηγηθεί καμία πολιτική συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι σε υπηρεσιακό απλώς επίπεδο ελήφθη η απόφαση αυτή. Δεν μας έχει δοθεί ακόμα μία επίσημη ανακοίνωση για την έκβαση της διαδικασία αυτής, αλλά δεδομένης πάντως της απόφασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν χωράει πλέον καμία αμφιβολία. Βρισκόμαστε σε ένα πλαίσιο που βλέπουμε ότι σε ότι όλο και περισσότερο λαμβάνονται αποφάσεις χωρίς να εμπλέκονται καθόλου οι κοινωνικοί εταίροι και ε, οι αποφάσεις αυτές επηρεάζουν τελικά το κοινωνικό μοντέλο για τα κράτη-μέλη και επηρεάζουν βέβαια πάρα πολύ τους εργαζομένους, ιδίως για τα κράτη-κοινά μέλη τα οποία υπόκεινται σε ένα μνημόνιο τη Τρόικα. Εφαρμόζονται δηλαδή όλο και περισσότερο μέτρα λιτότητας χωρίς να έχει προηγηθεί κανένας κοινωνικός διάλογος και βέβαια επηρεάζονται για αμοιβέ οι εργασιακές συνθήκες και το καθεξής. Ξέρετε ότι αυτό δεν συνδέεται απόλυτα με τον διεθνικό χαρακτήρα των διαπραγματεύσεων, αλλά απλώς σας υπενθυμίζω το όλο πλαίσιο στο οποίο λαμβάνει η χώρα αυτή η συζήτηση που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Επίσης, γίνεται μια στιγμή όπου βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μπλοκάρει όλα τα λεγόμενα κοινωνικά κείμενα. Η συνάδελφος Κορνέλισεν αναφέρθηκε στη δυνατότητα ένταξης της κοινωνικής διάταξης στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θέλει να δημιουργήσει μια πραγματική οικονομική και νομισμανική ένωση Ελπίζω να έχει δίκιο ο συναδελφό μας και όντω να προσθεθεί αυτή η κοινωνική διάσταση, γιατί εγώ αυτό το, αυτό το οποίο βλέπω επί του παρόντος είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επιτάπητο δύο έγγραφα, τα οποία ουσιαστικά μένουν πολύ περισσότερο στο ζήτημα της δημοσιονομικής πειθαρχία, το αν έχει να κάνει με τον προσυντονισμό των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και το άλλο έχει να κάνει με το νέο αυτό μέσο σύγκλησης για την ανταγωνιστικότητα, ενώ δεν λέγεται τίποτα και δεν υπάρχει κανένα κείμενο για το κοινωνικό μοντέλο, για την κοινωνική διάσταση. Τώρα, για ποιο λόγο τα λέω όλα αυτά. Τα λέω γιατί και εμείς φέρουμε μια κάποια ευθύνη. Στα διάφορα στάδια του κοινωνικού διαλόγου, όπως εξελίσσεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις έχουν διδραματίσει ένα κάποιο ρόλο γιατί η υλοποίηση των, εθνικών επιτροπών, των, συγγνώμη, των Ευρωπαϊκών Επιτροπών Εργαζομένων ουσιαστικά προσπαθούν να δημιουργήσουν μια κάποια δομή κοινωνικού διαλόγου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ξέρουμε ότι αυτές οι επιτροπές εργαζομένων λειτουργούν σχετικά καλά. Είναι αποτελεσματικές και αυτό το βλέπουμε για παράδειγμα σε κάποια σε επιχειρήσεις όπως η ArcelorMittal, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εργαζομένων προσπάθησε να αποφύγει το να στρέφεται μία χώρα ενάντια στην άλλη, χώρες δηλαδή στις οποίες ε, δραστηριοποιείται η επιχείρηση αυτή. Το ερώτημα όμως το οποίο τίθεται αυτή τη στιγμή είναι πώς θα καταφέρουμε να προασπιστούμε την κοινωνική διάσταση οικονομικής και νομισματικής ένωσης σε μακροοικονομικό επίπεδο και πώς θα καταφέρουμε να ανταποκριθούμε στο αίτημα αυτό, να υπάρχει ένας κοινωνικός διάλογος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Καταλαβαίνω αυτό το οποίο είπατε για την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων και όντω συμφωνώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Θα πρέπει όμως αυτή η αυτονομία των κοινωνικών εταίρων να προσαρμοστεί κάπως στην κατάσταση στην οποία αντιμετωπίζουμε. Αυτό το οποίο βλέπουμε επί του παρόντος είναι ότι ε, οι κοινωνικοί εταίροι στα πλαίσια ενός ε, μιας μακροοικονομικής ε, συζήτησης είναι πάρα πολύ περιορισμένος ο ρόλος τους. Και βλέπουμε πώς αντιμετωπίζονται πολύ συχνά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ο τρόπος με τον οποίο διδραματίζεται ο κοινωνικός διάλογος και ο τρόπος με τον οποίο συνάπτονται οι συμφωνίες ή εκτιλήσουν οι διαπραγματεύσει οι διεθνικέ ουσιαστικά παρουσιάζουν τα ίδια κάπως προβλήματα. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να φέρουμε το ένα επίπεδο εναντίον του άλλου. Και μπορούμε να διατηρήσουμε όντω την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων, αποτελέσει δηλαδή αυτό μια θεμελιώδη αρχή του μοντέλου που θα ακολουθήσουμε, αλλά από την άλλη, παράλληλα, θα πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί Πώ λειτουργούν οι κοινωνικοί εταίρες στην πράξη. Στη δική μα Επιτροπή έχουμε ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα. Βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προωθήσει την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων, αλλά αυτό οδήγησε στο να χάσουμε πέντε ολόκληρα χρόνια, ιδίω όσον αφορά την οδηγία για το χρόνο εργασία βλέπετε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καν νομοθέτημα κατά τη διάρκεια της δικής μας τουλάχιστον θητείας, γιατί είδαμε πώς λειτουργήσαν τελικά και οι κοινωνικοί εταίροι. Πέρα δηλαδή από την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων θα πρέπει να μπορεί και ο Ευρωπαίος νομοθέτης να λαμβάνει δράση, ιδίως όταν υπολείπονται των υποχρεώσεών τους οι κοινωνικοί εταίροι. Είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να τονίσουμε τα πλαίσια στα οποία διεξάγεται αυτή όλη η συζήτηση. Ποια είναι δηλαδή η παρούσα συγκυρία την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και να πω και κάτι ακόμα σε σχέση με αυτά που μας είπε και ο εισηγητής για, τον παγκόσμιο, για την Παγκόσμια Οργάνωση Εργασίας. Ξέρετε ότι ε, ο Αλεχάνδρο Φέρκας και ένας ακόμα συνάδελφος συμμετείχαν στην προηγούμενη συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και αυτό το οποίο μας έκανε πραγματικά εντύπωση είναι πόσο έχει μετατραπεί το πνεύμα εργασίας αυτού του οργανισμού μέσα σε πέντε χρόνια. Πριν από πέντε χρόνια η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας μας έλεγε ότι οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να λειτουργούν περισσότερο, να συμμορφωθούν περισσότερο με τις συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και να εφαρμόσουν τη σύμβαση αυτή εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ τώρα, πέντε χρόνια μετά, αυτό το οποίο μας είπανε είναι ότι είναι σημαντικό βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση να επικυρώσει τη σύμβαση αυτή γιατί αποτελεί πλέον τον ελάχιστο κοινό παρανομαστή του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Πρέπει λοιπόν να καταφέρουμε να δούμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτή τη σύμβαση της ε, Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και πώς θα καταφέρουμε να νομοθετήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο παράλληλα. Πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή να καλέσουμε και κάποιον εκπρόσωπο της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, προκειμένου να έχουμε πλέον με τον οργανισμό αυτό ένα πιο διαθρωμένο διάλογο και να καταφέρουμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τη σύμβαση αυτή, αυτού του οργανισμού, η οποία θα πρέπει να αποτελέσει βάση, όπως σας είπα. Αυτές οι παρατηρήσεις είχα να κάνω, δεν θα ήθελα να τις εκλάβετε ως απεσιόδοξες παρατηρήσεις, αυτό το οποίο θέλω είναι να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τον εισηγητή μας να είναι ιδιαίτερα φιλόδοξος, συγκεκριμένος και σαφής στην σύνταξη της έκθεσής του αυτή, αυτής και στα πλαίσια ενός περιβάλλοντος το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό. Δεν ξέρω αν θέλει κανείς άλλο το λόγο. Όχι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μήπως, ούτε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επομένως δίνω πάλι το λόγο στον εισηγητή μας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ήξερα ότι το θέμα θα ήταν δύσκολο, αλλά τόσο ακαθόδες δεν το έχω φανταστεί. Ήδη αρχίζει αυτό από τους ορισμούς που μπαίνουν σε αυτή τη συζήτηση και χρησιμοποιούνται. Μα δεν πρόκειται για διασυνοριακές συλλογικέ διαπραγματεύσεις για τους μισθούς, το είπαμε αυτό. Το είπε και ο κύριος Λούτβιξον και συμφωνώ απολύτως. Το λέω και στην έκθεσή μου. Οι συλλογικέ διαπραγματεύσεις είναι εθνικό θέμα και είναι και στα συντάγματα κατοχυρωμένο. Υπάρχει ένα εθνικό πλαίσιο, η ένωμη τάξη της κάθε χώρας. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν μπορούμε ούτε να το ζητήσουμε ούτε να το ρυθμίσουμε. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι συμφωνίες επιχειρήσεων μεταξύ τους με τα επιχειρησιακά συμβούλια, με την εκπροσώπηση των εργαζομένων, των συνδικάτων και είναι εταιρείε που έχουν ε, πολλά εργοστάσια στην Ευρώπη, τουλάχιστον δύο σε δύο χώρες. Και αυτά θα πρέπει να ρυθμίζονται. Βεβαίως θα πρέπει να συμφωνήσουμε ποιο θα είναι το νομικό πλαίσιο. Τουλάχιστον να συμφωνούν οι εταίροι για το ποιους εργαζομένους αφορά αυτό, γιατί και ακόμα και αυτό μπορεί να έχει διαφορά. Ας πούμε, στη Γερμανία το αντίστοιχο δίκαιο έχει άλλη ε, εμβέλεια ως προς το ποιους αφορά. Επίσης, σε άλλες χώρες θα πρέπει να λύθει το θέμα της εκπροσώπησης. Τα επιχειρησιακά συμβούλια δεν είναι παντού τα ίδια όπως στη Γερμανία, την Αυστρία ή αλλού. Πώς εκπροσωπούνται οι εργαζόμενοι και ποιος μπορεί να συναποφασίζει. Το άλλο είναι το θέμα της επέλυσης των διαφορών και των διακανονισμών. Και πάλι σε αυτή τη συζήτηση κινούμε από διαφορετικά επίπεδα. Δεν είναι μόνο το δικαίωμα στην απεργία. Είναι και όταν υπάρχει σύγκρουση στην υπογραφή αυτής της συμφωνίας, στο επίπεδο της επιχείρησης, ποιος το λύνει αυτό όταν κάποιος δεν τηρήσει αυτά που έχει υπογράψει ένα από τα δύο συμβαλόμενα μέρη. Δεν υπάρχει ένα τέτοιο πλαίσιο. Δεν μπορεί να προσφύγει ο άλλος κάπου. Και δεν θέλω εγώ να το αφήσουμε στα χέρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γράψτε ένα πλαίσιο. Εμείς θα πρέπει να βοηθήσουμε να αναπτυχθεί με προτάσεις δικές μας και με τους κοινωνικούς εταίρους να συνεννοηθούμε για να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο νομικό πλαίσιο. Εκκινούμε δηλαδή βοηθούμε σε μια διαδικασία βελτίωσης του ευρύτερου κοινωνικού διαλόγου. Και δεν θα πρέπει να κομπάζουμε ότι τα ξέρουμε καλύτερα από τους εργατολόγους ή από τα συνδικάτα. Αλλά χρειάζεται κάποια ρύθμιση, μας λείπει αυτή. Αυτό μας το είπαν στην ακρόαση οι επιρρογνώμονες. Και αυτό θέλω εγώ να χρησιμοποιήσω. Θα γίνει πραγματικά μια πολύ συναρπαστική συζήτηση. Ο καθένας έχει τις εμπειρίες του, ε, τις εθνικές και από τα διάφορα συστήματα συλλογικών συμβάσεων και στις χώρες και στα εργοστάσια και ακόμα και από τη θεώρηση των πραγμάτων. Τι γίνεται με το εργατικό δίκαιο, τι γίνεται με το δίκαιο των επιχειρήσεων, όλα αυτά είναι έκθεση πρωτοβουλία, είπαμε, και δεν υποθέτω ούτε θεωρώ ότι θα φτιάξουμε ένα συνταγματικό νόμο για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις στην Ευρώπη. Αλλιώς χάνουμε τελείως το στόχο μας. Αλλά μια συζήτηση μπορούμε να την αρχίσουμε. Και νομίζω και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδιαφέρεται γι' αυτό και πολλή δουλειά θα έχουμε, αλλά και ενδιαφέρουσα. Σα ευχαριστώ. Euh, Σας ευχαριστούμε λοιπόν. 7 Μαΐου η προθεσμία κατάθεση ε, τροπολογιών, 7 Μαΐου 12 το μεσημέρι. Θα εξετάσουμε τι τροπολογίε όταν συνεδριάσουμε στι 29 και 30 Μαΐου. Θα εξετάσουμε τι τις τροπολογίε στι 19 Ιουνίου και θα ψηφίσουμε στι 20 Ιουνίου και θα περάσει στην Ολομέλεια έκθεση αυτή το Σεπτέμβριο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώσαμε τις εργασίες μας και θα σας ξαναδώ στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας στις 7 Μαΐου στις 10 ώρα το πρωί.